Uh, welcome everybody. Καλώς ορίσατε. Καλημέρα σε όλους. Θα μιλήσω σου ειδικά. Καλώς ορίσατε λοιπόν και πάλι. Καλημέρα σε όλους. Ας συνεχίσουμε τις εργασίες μας μετά από την ε, χθεσινή μας δουλειά και τη χθεσινή μας συνεδρίαση. Θα εξετάσουμε το σημείο 10 της ημερήσιας διάταξης για τα δικαιώματα των γυναικών στις χώρες των Βαλκανίων που είναι υποπροσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν από αυτό όμως να καλωσορίσω την ομάδα επισκεπτών η οποία είναι σήμερα μαζί μας. Είναι 30 φοιτητές από το Μιλάνο προσκεκλημένοι της κυρίας Κώστα. Σας καλωσορίζουμε θερμά. Καλώς ήλθατε. Και έχουμε και επισκέπτες από την Επιστροπή για την προστασία των γυναικών και των παιδιών της ΑΣΕΑΝ, της Ένωσης Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας. 20 επισκέπτες από αυτή την Επιτροπή αυτής της οργάνωσης. Καλώς ήλθατε κι εσείς. Εσείς είστε η επικεφαλής της αντιπροσωπείας. Θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε και να σας δώσουμε το λόγο. Να σας πω ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να συνομιλήσουμε κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού διαλύματος. Καλώς ήρθατε κι εσείς, είστε ευπρόσδεκτοι στην ομάδα μας. Ας πάμε τώρα στο σημείο 10. Τα δικαιώματα των γυναικών στις υποψήφιες βαλκανικές χώρες. Να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, την κυρία Κορνέλησεν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. δεν είναι πολλοί σκιώδεις εισηγητές παρόντες σήμερα εδώ, δυστυχώς, αλλά ας ελπίσουμε ότι με τη μόνη σκιώδη εισηγήτρια που βρίσκεται εδώ μπορούμε να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω όλους για τις τροπολογίες που μου υποβάλατε. Πάνω από 100. Πολύ καλές. Οι μισές μάλιστα είναι και δικές μου. Αλλά όχι απολύτως δικές μου, όχι εντελώς δικές μου. Δηλαδή τι κάναμε, στείλαμε το σχέδιο έκθεσης σε πολλούς και διαφόρους, τουλάχιστον σε 100 μη κυβερνητικέ οργανώσεις, φορείς, εμπειρογνώμονες, πρέσβεις, ε, εκπροσώπους των, των κρατών στις υποψήφιες βαλκανικές χώρες και μας έστειλαν feedback με διάφορες υποδείξεις, κάποιες από τις οποίες ενσωματώσαμε και ενστερνιστήκαμε. Οι 50 τροπολογίες λοιπόν από τις 100 είναι το προϊόν της συνεισφοράς των συνομιλητών μας στις χώρες αυτές καθεαυτές. Πράγμα που σημαίνει ότι ήδη η συζήτηση ε, που εξελίσσεται στις χώρες αυτές είναι πολύ ζωντανή με αντικείμενο την έκθεση. Και αυτό είναι άλλωστε και ένας από τους βασικούς μας στόχους. Ένας από τους στόχους της έκθεσης έχει ήδη επιτευχθεί πριν από την ψήφισή της, ε, διότι στόχος μας είναι η ενθάρρυνση και η ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών στις υποπροσχώρηση χώρες. Οι τροπολογίες των μελών συμπεριλαμβάνουν πολλά θετικά στοιχεία που συμπεριλήφθηκαν στο σχέδιο της έκθεσης, εν μέρη και γιατί δεν είμαι από Πολύτο ειδικό ειδική σε αυτό το τομέα και εν μέρη διότι πάντοτε μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει πολλές και διαφορετικές διατυπώσεις σε ένα σχέδιο έκθεσης. Θέλω να ευχαριστήσω το μέλος, ε, την κυρία Βάλτρο, η οποία βοήθησε στη σύνταξη της ε, τροπολογίας για τις γυναίκες Ρωμά. Να ευχαριστήσω τα μέλη που ε, μίλησαν για το ψήφισμα 1325 για την, το επιχειρηματικό πνεύμα. Να ευχαριστήσω την κυρία Ιντβέλτ, η οποία έβαλε τα αντισυλληπτικά στην έκθεση. Και αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Κάποια σημεία μένει να συζητηθούν. Π.χ. οι ποσοστώσεις των γυναικών στην πολιτική ζωή. Γνωρίζω ότι οι απόψεις διήστανται από αυτού. Στην έκθεση αυτό το οποίο λέμε είναι ότι Δεν καλούμε τόσο τις χώρες να επιβάλλουν ποσοστώσεις για τη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική ζωή, αλλά λέμε ότι εάν οι χώρες έχουν επιλέξει να θεσμοθετήσουν ποσοστώσεις, τότε θα πρέπει αυτές να τις τηρούν. Δεν είναι δικιά μας δουλειά ως Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχουμε κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα αυτό. Ε, Επομένω, δεν ε, νομιμοποιούμεθα ε, να καλέσουμε τις χώρες να εδραιώσουν ποσοστώσεις όταν δεν υπάρχουν στη συγκεκριμένη χώρα. Αυτό όμως το οποίο τις καλούμε να κάνουμε είναι να τις, εφαρμόσεις, αν τις, να τις εφαρμόσουν αν τις έχουν υιοθετήσει. Ένα άλλο πολιτικό ζήτημα είναι το πώς θα αποκαλείται η Μακεδονία, λέει ο Μιλήτρια. Η κυρία Γιανακουδάκη πρότεινε να γράψουμε όλη την ονομασία, την πλήρη. Η κυρία Παπαδοπούλου πρότεινε να χρησιμοποιήσουμε τη συντομογραφία, το φύρομ δηλαδή. Εγώ προσπάθησα να είμαι κάπως πρωτότυπη. Σύντμησα τις πρώτες τρεις λέξεις, αλλά όχι την τελευταία. Φύρο Μακεδονία. Σαν συμβιβαστική λύση. Βεβαίως, εναπόκειται στον καθένα από τη δική του, αναλόγως με τη δική του πολιτική σκοπιά, να ψηφίσει υπέρ της μίας οποιασδήποτε εκ των τριών ε, δυνατοτήτων. Βεβαίως θα λυπούμουν πολύ αν δεν θα επιτρεπόταν να χρησιμοποιηθεί και το επίθετο «μακεδονικός». Ο κανόνας είναι ότι όσο ουσιαστικό όταν αναφερόμαστε στη χώρα λέμε πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, αλλά μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ως επίθετο και να πούμε η μακεδονική κυβέρνηση. Επομένως ο καθένας έχει την επιλογή αναλόγως με την πολιτική του ομάδα. Τώρα, επί του περιεχομένου, κάτι το οποίο θα εξετάσω πιο επισταμένος. Ως προς την Αλβανία ζητούμε ε, ξεχωριστό επίτροπο για την ισότητα των φύλων, διότι ε, ε, εκεί θα μπορούν να υποβάλλονται εκθέσεις, αναφορές μάλλον, από γυναίκες που έχουν υποστεί διακρίσεις. Οι αλβανικές μη κυβερνητικές οργανώσεις μας είπαν ότι αυτό θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο. Από την άλλη, ε, άλλοι λένε ότι είναι ένας επιπρόσθετος θεσμός, ένα επιπρόσθετο θεσμικό όργανο που συστήνεται και αυτό ίσως ήταν, είναι κάπως δίσκαμπτο. Ε, θα το συζητήσουμε να δούμε ποιος είναι ο κατάλληλος τρόπος, ο καλύτερος τρόπος να προχωρήσουμε. Κατά τα λοιπά θα είναι εύκολο να καταλήξουμε σε κάποιες επικοδομητικές συμβιβαστικές λύσεις. Κατά τη διάρκεια της Συνόδου της Ολομέλειας στο Στρασβούργο τον Μάρτιο θα προσπαθήσω να οργανώσω μία συνάντηση με τους κοιόδης εισηγητές. Την πρώτη φορά που συζητήσαμε την έκθεση αυτή υποβλήθηκε ένα επιχείρημα σε σχέση με την Κροατία. Ότι δηλαδή στο σχέδιο έκθεσης μου καλώ την Κροατία να προσαρμόσει περισσότερη από την νομοθεσία της το ευρωπαϊκό κεκτημένο σε κάποιους από τους τομείς που έχουν να κάνουν με την ισότητα των φύλων. Από ό,τι μου λένε το έχει ήδη κάνει αυτό η Κροατία. Επομένως το επιχείρημα αυτό η σχετική διατύπωση μπορεί να διαγραφεί από την τελική έκθεση. Και τέλος να επισημάνω ότι στο στάδιο της Ολομέλειας, της ψήφισης στην Ολομέλεια, μπορεί ο εισηγητής να τροποποιήσει την έκθεση με προφορικές τροπολογίες ε, προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, εάν προκύψουν νέα στοιχεία που καθιστούν κάποια τέτοια τροποποίηση απαραίτητη. Το καλύτερο θα ήταν να καταφέρουμε να διαγράψουμε το περιεχόμενο της μισής έκθεσης ούτως ή άλλως. Ήδη, διότι τα κράτη έχουν κάνει πολλά και τα δικαιώματα των γυναικών τη χάνουν καλύτερης προστασίας σε αυτές τις χώρες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ η κυρία Νεβιτάλοβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν είμαι σκιώδης εισηγήτρια η κυρία Ότσο Κλέβα είναι η σκιώδη εισηγήτρια και θα διαβάσω την τοποθέτησή τη. Σα ευχαριστώ για την έκθεσή σα. Είναι πολύ σημαντική η έκθεση αυτή. Εφιστά την προσοχή στο πρόβλημα των δικαιωμάτων των γυναικών και υπάρχει ελπίδα ότι θα ενισχύσει την ισότητα των φύλων στην περιοχή. Οι Βαλκανικές χώρες έχουν σημειώσει πρόοδο στον τομέα της ισότητας των φύλων και θα πρέπει να τη συγχαρούμε, ειδικότερα την Κροατία, διότι έχει ευθυγραμμίσει στη μεγαλύτερη της πλειονότητα την νομοθεσία της με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Εν τούτης, πολλά μένουν να γίνουν. Οι τροπολογίες της κυρίας Κλέβα ε, κοφκιούς για τα διάφορα θέματα. Θέση της γυναίκας στην αγορά εργασίας συνεχίζουν να παίρνουν χαμηλότερους μισθούς. Θα πρέπει να αυξηθεί η πρόσβασή τους στην εργασία γενικότερα και στην αγορά για να ανισχυθεί και το εισόδημά τους. Θα πρέπει οι κυβερνήσεις να έχουν μέτρα για ίσες ευκαιρίες για να μειωθεί η μισθολογική ανισότητα. Αυτό οδηγεί και σε διαφορές στις συντάξεις και συνταξιδοτικό κενό και τελικά οι γυναίκες στο τελευταίο στάδιο της ζωής τους είναι σε κατάσταση ακόμα μεγαλύτερης φτώχειας. Και τέλος ε, ε, υποεκπροσωπούνται οι γυναίκες στην πολιτική σκηνή, στο πολιτικό στερέωμα. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τις Βαλκανικές χώρες αλλά και για την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξού και η ποσόστοση και η τήρηση της ποσόστοσης χρειάζεται να εδραιωθεί και να εφαρμοστεί και θα πρέπει να συνοδεύεται από αποτελεσματικές νομικές κυρώσεις. Τέλος, θα πρέπει να βρεθούν λύσεις για τις σκληρά εργαζόμενες γυναίκες που δυσκολεύονται να συμφιλειώσουν επαγγελματική και προσωπική οικογενειακή ζωή και θα πρέπει να υπάρξουν περισσότερες εκστρατείες συνειδητοποίηση καταπολεμώντας τα στερεότυπα και τις διακρίσεις. Στερεότυπα και διακρίσεις που είναι βαθιά ριζωμένα στην παράδοση των υποψήφιων βαλκανικών χωρών. Και μάλιστα οι Γυναίκε Ρωμά ε, υπόκεινται, υφίστανται διπλέ διακρίσει και θα πρέπει να υπάρξει ένα πλαίσιο των διακρίσεων ώστε να αγγιόμαστε τα δικαιώματα των γυναικών αυτών. Τέλο, για να προωθήσουμε την ατζέντα μα για την ισότητα των φύλων στα Βαλκάνια θα πρέπει να έχουμε πολιτικέ mainstreaming τη διάσταση του φύλου. Οι κυβερνήσει πρέπει να ενισχύσουν τη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική να έχουν καλύτερη πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην υγεία. Θα πρέπει οι δεσμεύσεις ε, να εφαρμοστούν στην πράξη. Η κυρία Κλέβα θέλει να ευχαριστήσει την εισηγήτρια για άλλη μια φορά για τη δουλειά που έχει κάνει και αδειμονεί για περαιτέρω συνεργαστία. Ευχαριστώ πολύ. Και ένα σχόλιο για το Φύρομ και το Μακεδονικό. Είναι προσωπικό μου σχόλιο, όχι σχόλιο της και όλες εισηγήτρες από πλευρά Εμένα μου αρέσει πολύ ο λαός αυτός. Έχω πολλούς ε, φίλους εκεί, αλλά θα πρέπει να σεβόμαστε ε, την ορολογία των Ηνωμένων Εθνών που είναι η επίσημη. Επίσημη ονομασία είναι το ΦΥΡΟΜ. Δεν μου αρέσει ούτε μένα, προτιμώ το Μακεδονία, αλλά αυτό είναι θέμα σκιώδου εισηγητής, εκείνη θα αποφασίσει γι' αυτό η σκιώδης εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις. Θέλει κάποιος άλλος το λόγο. Ιδάλλως, ας μας πει ο, ο πρόσωπος της Επιτροπής, ο κ. Σόπτεμπακ, αν θέλει να παρέμβει. Υπάρχει κάποιος από την Επιτροπή. Είμαι η κυρία Σάντλε από τη Γενική Διεύθυνση Διεύρυνσης. Νομίζω ήδη γραπτώς επικοινωνήσαμε για τις τροπολογίες με την συγκεκριά. Και με χαρά είδαμε ότι υπάρχει τόσο ενδιαφέρον με τις τροπολογίες. Πραγματικά αυτό μας ικανοποιεί. Επίσης, τα σχόλια που κάναμε στον πρώτο γύρο των συζητήσεων έχουν συμπεριληφθεί κατά μεγάλο μέρος, ενώ η συγγήτρια έχει καλύψει και υπέρ το δέον κάποιες φορές αυτά που η Επιτροπή έχει αναφέρει σε δικές της εκθέσεις για τις χώρες αυτές, το περασμένο φθινόπωρο κιόλα. Έχουμε ακόμη κάποια σχόλια, τα οποία ήδη έχουμε μεταβιβάσει στην εισηγήτρια και επίσης η νομική ευθυγράμμιση εντωμεταξύ έχει ολοκληρωθεί στην Κροατία σε αυτό το τομέα. Δεν χρειάζεται λοιπόν πλέον να το θεωρούμε ζήτημα και να αναφέρεται και στην έκθεση. Επίσης, όσον αφορά την Κροατία και πάλι, η τροπολογία 69 καλεί την κροατική κυβέρνηση να προσφέρει δωρεάν νομική βοήθεια σε θύματα διακριτικής μεταχείρισης και διακριτικών συμπεριφορών. Καλύτερη διατύπωση θα ήταν να βελτιώσει την πρόσβαση στην νομική αρρωγή, την δωρεάν νομική αρρωγή. Έχουμε παρατηρήσει σε πολλές περιπτώσεις ότι το να λάβει ήδη κανεί την δωρεάν νομική αρρωγή είναι πολύ περίπλοκο. Οι κροατικέ αρχέ αυτή τη στιγμή ακριβώ προσπαθούν να μεταρρυθμίσουν τη σχετική νομοθεσία για την δωρεάν νομική αρρωγή και προκειμένου να υπάρχει ευκολότερη πρόσβαση για όλου. Σε ό,τι αφορά το κοσυφοπαίδιο, είχαμε ένα σχόλιο για την τροπολογία 76, όπου καλείται η κυβέρνηση του κοσυφοπαιδίου να απευθυνθεί στο Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων. Δεν έχουμε αντίρρηση ως προς την αυτή καθεαυτή. Όμως, ας σημειώσουμε ότι αν πρέπει να έρθει σε επαφή το ίδιο, η ίδια υπηρεσία του Πρωθυπουργού, με το, οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού με το Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, αυτό δεν είναι αναγκαίως η καλύτερη επιλογή.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 Yeah, Mrs. Kleva, I think I'm uh, I'm going to recommend a plus for for almost all her amendments. Uh, They were very valuable um, uh, contributions. Νομίζω λοιπόν ότι η κριτική μεταχείριση κατά των γυναικών Ρωμά είναι ένα σημαντικό θέμα. Εγώ ήδη μιλώ για την διτή διακριτική μεταχείριση γυναικών που ανήκουν και στην ομάδα των λεσβιών, ομοφιλοφίλων και ούτω καθεξής. Στις περισσότερες από τις χώρες ε, των Βαλκανίων που βρίσκονται στη δικασία της ε, προσχώρησης. Χαίρομαι που μπορούμε να επενέσουμε αυτές τις χώρες και για πολλά χαρακτηριστικά τους. Αυτό δείχνει ότι τα περασμένα χρόνια στη διαδικασία της προσχώρησης πολλά άλλαξαν και βελτιώθηκαν ήδη βλέπει κανείς ότι, ότι η Κροατία λόγου χάρη είναι στα πρόθυρα της ε, προσχώρησης. Και μάλιστα θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως παραδείγμα για τις υπόλοιπες χώρες. Ιδίω η υπεύθυνη διαμεσολαβήτρια, η ombudswoman για τα ισότητα των φίλων είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Για την πρώην Μακεδονία πολλά έχουν υποθεί. Εγώ Απλώ δεν ήθελα να χρησιμοποιήσω ολόκληρη τη διατύπωση πρώην και Δημοκρατία τη Μακεδονία ή Φύρομ. Δεν ήθελα να ε, λάβω θέση. Το να χρησιμοποιήσω την επίσημη ονομασία όπως αναφέρεται από τον ΟΗΕ είναι και αυτό ουσιαστικά σαν να ρολευτεί Ήθελα λοιπόν από τη δική μου την πλευρά να βρω ένα τρόπο να μην τοποθετηθώ και να σεβαστώ και τα αισθήματα των ίδιων των ε, Μακεδόνων. Είναι όμως πολιτική επιλογή του καθενός. Ίσως εδώ απλώς να μην δώσω μια κατεύθυνση για την ψηφοφορία. Είναι μια ελεύθερη επιλογή για τον καθένα. Για τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. για την τροπολογία 69 για την δωρεάν νομική αρρωγή στην Κροατία. Θα προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε αυτό με μια προφορική τροπολογία ή να δούμε κατά πόσον με τις συμβαστικές λύσεις κάπως μπορούμε να το καλύψουμε. Ενώ για το κοσυφοπαίδιο το να τεθεί αυτό υπό την αγίδα ε, του Πρωθυπουργού είναι κάτι που εντάξει θα μας δώσει την εντύπωση ότι η κυβέρνηση δείχνει πραγματική βούληση να αναλάβει δράση, αλλά δεν μπορεί να τα αναλαμβάνει και η υπηρεσία του Πρωθυπουργού. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την ουδετερότητα και την αμεροληψία. Θα πρέπει να βρεθεί μια μέση οδός για να λειτουργήσει αποτελεσματικά αυτή η συνεργασία με την απαραίτητη αφοσίωση και την ανεξαρτησία που είναι απαραίτητη. Αναμένω τώρα τη συζήτηση για τι συμβαστικέ τροπολογίε και είμαι βέβαιη ότι θα καταλήξουμε σε μια πολύ ικανοποιητική έκθεση. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Και να σας δώσω τώρα το χρονοδιάγραμμα για το θέμα αυτό. Η Επιτροπή μας θα ψηφίσει στις 20 Μαρτίου. Και η Ολομέλεια μάλλον θα το συζητήσει τον Μάιο. Ας προχωρήσουμε. Ευρωπαϊκό Ταμείο ενίσχυση των Απόρων. Να δώσω και πάλι το λόγο στην εισηγητρία που για άλλη μια φορά είναι η κυρία Κορνέλισεν. Μάλιστα. Το Ταμείο για τους Απόρους λοιπόν. Έχουμε μια γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης. Και λέμε ότι το ταμείο αυτό είναι ένα ταμείο γυναικών στην ουσία. Οι γυναίκες έχουν πολύ μεγάλη εκπροσώπηση ανάμεσα στους απόρους, διότι τις τελευταίες δεκαετίες δεν έχει λυθεί το πρόβλημα της, ε, το... της γυναικείας φτώχειας. Η φτώχεια έχει πλέον γυναικείο πρόσωπο. Ακόμα και τώρα, οι γυναίκε σε μια οικογένεια, σε ένα νοικοκυριό είναι εκείνες που αγοράζουν το φαγητό, που μαγειρεύουν, εκείνες που φροντίζουν για τον επιστημισμό της, ε, της οικογένειάς τους και η μείωση στο εισόδημα πλήττει εκείνες και γίνεται αντιληπτή από αυτές στην αρχή. Τι έκανα στη γνωμοδότηση, προσπάθησα να δώσω έμφαση στους εξαρτώμενους ανθρώπους, κυρίως τις γυναίκες, και στα προγράμματα που είχαμε τα τελευταία χρόνια, το πλεόνασμα τροφίμων δινόταν στις ε, τράπεζες φαγητού ή στα συσίτια για τους απόρους. και προτείνω να συνεχιστεί αυτό. Υπήρξε μία μειοψηφία στο Συμβουλίο η οποία μπλόκαρε την ε, ύπαρξη του ταμείου αυτού, την απελευθέρωση κονδυλίων για αυτό το ταμείο και έτσι τα κονδύλια τώρα είναι λιγότερα από ό,τι στα προηγούμενα προγράμματα. Φαίνεται σαν, το, σαν η αντίδραση αυτή του Συμβουλίου και η αντίστασή του να έχει επιληθεί το Ταμείο για τους Απόρους συμπεριλήφθηκε τώρα στα πλαίσια του νέου δημοσιονομικού, δημοσιονομικού πλαισίου και θα έχει λοιπόν τα κονδύλια. Αυτό όμως δεν λύνει το πρόβλημα ότι πλέον τα κονδύλια είναι λιγότερα από ό,τι ήταν παλαιότερα. Και να πω επίση ότι όλε οι χώρε είναι υποχρεωμένε να συμμετάσχουν σε αυτό. Υπάρχουν χώρε όπω το Ηνωμένο Βασίλειο, όπω η Γερμανία, η Σουηδία επίση και οι κάτω χώρε οι οποίες θα αναγκαστούν να συμμετέχουν ακόμα και αν δεν το επιθυμούν και αυτές οι χώρες θα πάρουν χρήματα από αυτό το ταμείο και έτσι θα υπάρχουν ακόμα λιγότερα χρήματα για να διαμοιραστούν στους υπόλοιπους. Εάν το ταμείο, εάν τα κονδύλια δεν αυξηθούν, τότε θα έχουμε πρόβλημα. Το ταμείο αυτό το χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο γυναίκες. Και κύριο μέλημά μας θα πρέπει να είναι η αποφυγή δημιουργίας περισσότερων εξαρτώμενων γυναικών. Επίσης, πιστεύω ότι είναι αρκετά σημαντικό να προσπαθήσουμε να δώσουμε στους οργανισμούς αυτούς της Τράπεζας Τροφίμων στα συσίτια τα μέσα για να προμηθεύονται τα ίδια τα τρόφιμα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, τον, ε, υπάρχουν πολλοί τόνοι ε, τροφίμων που πετιούνται στα σκουπίδια κάθε χρόνο. 90 εκατομμύρια τόνοι. Και αυτό θα μπορούσε να δοθεί στους οργανισμούς αυτούς αυτές οι τράπεζες τροφίμων θα μπορούσαν να έχουν καλύτερη πρόσβαση σε τρόφιμα εάν είχαν τα μέσα. Χρειάζεται συνειδητοποίηση του κοινού. και διευκόλυνσή τους με διάφορα μέσα έτσι ώστε να μπορέσουν να έχουν αυτή την πρόσβαση. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να φροντίσουμε για αυτό, έτσι ώστε οι γυναίκες που εξαρτώνται από αυτά τα μέσα να μπορέσουν να θρέψουν τις οικογένειές τους. Και αυτό είναι το σχέδιο μέχρι το 2014. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Κώστα, η οποία ζήτησε πρώτο το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εξαιρετική της δουλειά τη γνωμοδότηση αυτή. Συμφωνώ ότι πρέπει να μιλήσουμε για ένδια και καταπολέμηση τη ένδια και μέσω αυτού του ταμείου που αντικαθιστά το προηγούμενο. Το προηγούμενο το οποίο ε, στηριζόταν και από την γεωργική πολιτική. Κάτι που πλέον θα καλύπτεται, πλέον, ε, θα καλύπτεται πλήρως από το σκέλος ε, της κοινωνικής πολιτικής. Πρόκειται για ένα στόχο που θα πρέπει να δώσει έμφαση στην προστασία των γυναικών. Εδώ πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Αν το ποσοστό της ένδυας ε, στην Ευρώπη με πάνω από 100 εκατομμύρια πολιτών στην Ευρώπη, το 1 τρίτο σχεδόν, ε, και οικογένειες ολόκληρες, παιδιά, ε, δυσκολίες πρόσβασης στα τρόφιμα, γυναίκες μόνες, ηλικιωμένες ή πολλές οικογένειες μονογονικές, βλέπουμε ότι όταν μιλάμε για φτώχεια δεν μιλάμε για κάτι ουδέτερο ή αδιάφορο. Γι' αυτό έχει δίκιο, έχει δίκιο ο συνάδελφο. Οι τροπολογίε που φαίνονται να μα απομακρύνουν από το θέμα το συγκεκριμένων των γυναικών στην πραγματικότητα είναι πολύ εύστοχες. Γιατί ακριβώς οι επιπτώσεις αφορούν κυρίω τι γυναίκε. Δεύτερη παρατήρηση. Θεωρώ και προσωπικώ σα με την πρόταση να είναι προαιρετική η συμμετοχή στο Ταμείο μέσω των μέλων. Ιδάλλως θα καταλήγαμε σε ένα παράλογο, σε μια παράλογη κατάσταση. Η, ο στόχος της καταπολέμησης της φτώχειας ως το 2020 για την επόμενη επταετία θα ερχόταν σε αντίφαση με, την, ε, με τις δραστικές περικοπές στο ταμείο αυτό 2,5 εκατομμύρια για 19 χώρε, 2,1 στην πρόταση του Συμβουλίου μάλιστα, για 28 χώρε σε σχέση με τι 19 που υπήρχαν πριν. Και με πάνω από 3 εκατομμύρια. Εδώ λοιπόν αυτό δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, ακόμη και σε χώρε που δεν είχαν ε, τέτοιε αναταραχέ ω τώρα. Επίση, να συμφωνήσω ότι θα πρέπει να υπάρχει διαφορετικό ποσοστό κάθε φορά, όπω προτείνει η εισηγήτρια. Η συμμετοχή κατά 5% είναι σημαντική, αλλά δεν μπορεί να είναι ομογενοποιημένο στοιχείο. Θα πρέπει ανάλογα με δείκτε να υπάρχουν διαφορέ αναχώρε και σωστά αναφέρεται και το θέμα τη προσοχή και των στατιστικών, των μη επεξεργασμένων στατιστικών ανά ηλικιακή ομάδα και ε, σε βάση οικογενειών. Όπω είπε η κυρία Κορνέλισεν, ο στόχο του νέου ταμείου, τη νέα φιλοσοφία του ταμείου, θα πρέπει να έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά διαφορετικά μεταξύ τους. Πρώτον, να μειωθεί η εξάρτηση ε, χωρίς να μιλάμε όμως για την ε, εξάρτηση φορέων ή ατόμων που δεν θα πρέπει να στηρίζονται καθόλου. Θα πρέπει με άλλα φορολογικά ή πολιτικά μέσα να τους στηρίξουμε. Κάποιος λέει λόγω χάρη μείωση του ΦΠΑ για όσους προσφέρει κοινωνικές παροχές ή μπορεί να στηρίζει τη διατροφική αλυσίδα με διαφορετικές τιμές. Συμφωνώ σε αυτό. Θα μπορούσαμε να στηρίξουμε την δημιουργία δικτύων δικτύων όπω στη χώρα μου που λειτουργήσαν και λειτουργούν ακόμα, που φέρουν πιο κοντά τους παραγωγούς τροφίμων στους καταναλωτές. Αυτό ονομάζεται στην Ιταλία κιλόμετρο τζέρο, 0 χιλιόμετρα, δηλαδή μείωση τη απόσταση μεταξύ του παραγωγού και του τελικού καταναλωτή. Αλλά κυρίω προβλέποντας στις επιστημιστικές παρεμβάσεις που θα πρέπει να προστατευτούν, να υπάρχουν και συνοδευτικά μέτρα, μέτρα υποστήριξη, τα οποία να μπορούν να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά τη φτώχεια. Νομίζω πρόκληση για το νέο ταμείο είναι να ακολουθήσει μια συνολική προσέγγιση για την καταπολέμηση ακριβώ τη ένδυα και του κοινωνικού αποκλεισμού. Νομίζω πάντω ότι σαφώ και έχοντα υπόψη ότι κάποιε κοινωνικέ πολιτικέ, ακόμη και το κοινωνικό ταμείο, δυστυχώ δεν επιτυγχάνουν του πραγματικού στόχου, θα πρέπει να σταθούμε σε αυτό και να σκεφτούμε ποια είναι η ουσία του ταμείου αυτού. Ότι θα πρέπει να είναι να το δούμε σε ένα όργανο που ήταν για τον ώρα ενδεικτικό. Όχι ανεπαρκέ, αλλά ενδεικτικό. Την πραγματική φτώχεια, τον πραγματικό αποκλεισμό δεν τον καταπολεμήσαμε. Απλώ τον αναχαιτήσαμε. Διαφορετική λοιπόν προσέγγιση, συνολικότερη, σφαιρικότερη, όχι μόνο με αυτό το ταμείο, αλλά θα πρέπει να αρχίσουμε να το μελετούμε να δούμε το ελάχιστο εισόδημα των πολιτών λόγω χάρη. Κάτι άλλο θα πρέπει η Ένωση μας ενδεχομένω να επεξεργαστεί για το μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Πάουελ έχει το λόγο. Μπάουερ. Ευχαριστώ πολύ. Φαίνεται ότι τώρα είναι το πρωινό της κυρίας Κορνέλης. Εν συγχαρητήρια λοιπόν για τη σκληρή σας δουλειά να προσθέσω κάποια πράγματα, κάποια σχόλια για την έκθεση αυτή. Καταρχάς μου φαίνεται μια σταγόνα στον ωκεανό η έκθεση αυτή, διότι το δίκτυο κοινωνικής πρόνοιας είναι τεράστιο και τα κονδύλια αυτά είναι πολύ λίγα. Η μείωση της φτώχειας δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσω αυτού του ταμείου, διότι αυτό το ταμείο έχει δημιουργηθεί για την ακραία φτώχεια και όχι για την φτώχεια γενικά. Θα μπορούσαμε να, πιστεύω πως θα μπορούσε τώρα να δημιουργηθεί μια νέα ομάδα εξαρτημένων ατόμων από αυτό το ταμείο. Αλλά ίσως αυτό είναι λίγο υπερβολικό. Σε γενικές γραμμές πάντως συμφωνώ με τη γνωμοδότηση, εκτός από ορισμένα σημεία, από ορισμένες τροπολογίες, την 30 συγκεκριμένα. βλέπω πως υπάρχουν διαφορετικά όρια όσον αφορά την πρόσβαση σε αυτά τα ταμεία και αυτό δεν το θεωρώ καλή ιδέα. σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, διότι η πρόσβαση σε αυτό είναι ανοιχτή για όλες τις χώρες. Δεν περιορίζεται η πρόσβαση σε ορισμένες, στις πιο φτωχές χώρες και αυτό πιστεύω πως αυτό θα έπρεπε να το συζητήσουμε περισσότερο. Δεν είμαι και πολύ υπέρ αυτού. Μετά, δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά τις ανακοινώσεις της Επιτροπής, αλλά πιστεύω ότι αυτές εστιάζονται πάρα πολύ στην επιστημιστική βοήθεια. Περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Γνωρίζουμε ότι η καταπολέμηση της φτώχειας γίνεται και μέσω της στέγασης, αλλά αυτό δεν το βλέπω να αναφέρεται πουθενά. Τι γίνεται με τη στέγαση. Και ιδιαίτερα αν δούμε και τις ε, μεγάλες χώρες, θα δούμε ότι το ταμείο αυτό, τα κονδύλια του ταμείου δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών όλων των κρατών μελών. Ε, τώρα, συμφωνώ με την κυρία Κονέλσεν στο ότι πρέπει να προσέξουμε και τους άλλους ε, οργανισμούς της Τράπεζας Τροφίμων, να δούμε εκείνες τι κάνουν και πώς προσπαθούν να βρουν και άλλους ε, και άλλες πηγές ε, κονδυλίων και όχι μόνο αυτό το ταμείο. θα μπορούσαμε ίσως να χρησιμοποιήσουμε αυτό το ταμείο και για κοινωνική στέγαση, αλλά εάν όχι, να ξανασκεφτούμε και να δούμε αν υπάρχει πιθανότητα έστω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Μονίτσα, Τσατέρ έχει το λόγο τώρα για την πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτριά μας, την κυρία Κορνέλισεν, για όλη τη δουλειά που έχει επιτελέσει σε αυτό το θέμα που μας ενδιαφέρει τα μάλα όλους και όλες, σε ένα θέμα το οποίο προσυπογράφουμε όλοι και όλες ανεξαρτήτως πολιτικής ομάδας. Όπως είπε και η κυρία Μπάουερ μόλις τώρα, ε, βρισκόμαστε σε σημείο κρίσιμο, σε μια καμπή, διότι η κρίση οξύνει την κατάσταση απόλυτης ένδυας και αυτή τη στιγμή με αυτό το ταμείο πρέπει να εξυπηρετήσουμε και την επισητιστική βοήθεια, αλλά και άλλες πολύ μεγάλες ανάγκες, δραματικές ανάγκες θα έλεγα, που αυθρίζονται στις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν στο πλαίσιο της επιστημιστικής βοήθειας. Αυτό λοιπόν το Ταμείο θα πρέπει να καταπολεμήσει την κατάσταση απόλυτης ένδυας, με ό,τι αυτό περιλαμβάνει, όλες τις, τις συνιστώσεις, και γι' αυτό το λόγο, όπως είπε και η κυρία Μπάουερ, θα ήθελα να επιμείνουμε σε αυτή τη διαφοροποίηση των δράσεών μας. Γνωρίζω ότι οι τράπεζες τροφίμων, τα εστιατόρια της καρδιάς όπως τα αποκαλούμε, οι οργανισμοί δηλαδή ε, που προσφέρουν φαγητό με οργανωμένο τρόπο, οι οργανισμοί που βοηθούν για τη στέγαση, για την πρόσβαση σε συνθήκες υγιεινής, που προσφέρουν συμβουλές ε, για τη διατροφή, ε, προσφέρουν συμβουλές ακόμα και για τη διαχείριση του πολύ μικρού προϋπολογισμού που μπορούν να έχουν οι άνθρωποι που το χρειάζονται. Πρέπει να στηριχθούν, η βοήθεια είναι πολλαπλή και θα πρέπει να συνεχιστεί. Θα ήταν άδικο να κλείσουμε τους ορίζοντες και να ε, περιοριστούμε μόνο στην ε, επισητιστική βοήθεια. Γνωρίζω ότι στην Ευρώπη αυτό είναι το κύριο θέμα. Θα πρέπει όμως να ανοίξουμε και άλλους διάβλους ε, και να εξερευνήσουμε και άλλα εδάφη σε αυτό τον αγώνα καταπολέμησης της απόλυτης ένδυας. Είπε η κυρία Κορνέλισεν ότι στην τελική είναι ένα ταμείο για τις γυναίκες. Γνωρίζω ότι εδώ είναι η Επιτροπή για τις γυναίκες. Θα ήταν σφάλμα όμως να περιορίσουμε τον ορίζοντά μας λέγοντας ότι πρόκειται για ένα ταμείο για τις γυναίκες, κύριε Πρόεδρε. Αυτό πιστεύω. Γνωρίζω και γνωρίζετε όλοι και όλες ότι έχουμε και ζητούμε ακόμα περισσότερες στατιστικές αναφύλο. Και αυτό είναι σωστό πρέπει να αναδείξουμε τη σημασία που έχουν οι γυναίκες. Οι, μονογονε... οι γυναίκες που είναι επικεφαλής σε μονογονεϊκή οικογένεια ε, και ούτω καθεξής. Συμφωνώ και τα στηρίζω όλα αυτά και συμφωνώ με το αίτημά σας για την ύπαρξη στατιστικών αναφύλων. Αυτό ναι, αλλά από εκεί μέχρι, και να... μέχρι το να πούμε ότι είναι ένα ταμείο μόνο για τις γυναίκες ή ένα ταμείο για τις γυναίκες η απόσταση είναι μεγάλη. Ουσιαστικά περιορίζουμε τους ορίζοντές μας και αποκόπτουμε τις γυναίκες από την κοινωνική διαφορετική πραγματικότητα μέσα στην οποία εντάσσονται. Ε, ζητώ συγγνώμη ενδεχομένως γιατί ε, τα λόγια μου είναι έτσι πολύ ε, έντονα αλλά είναι ένα θέμα που με απασχολεί ιδιαιτέρως. Καλό είναι να ζητήσουμε να υπάρχουν συστατιστικές και να πληθυσμιακή ομάδα. Αυτό το οποίο διαπιστώνω σήμερα είναι το εξής. Έχουμε διαφορετικές ανάγκες που πρέπει να καλύψουμε. Ανάγκη για στέγαση, για ένδυση, για σύτηση. Και όλες αυτές οι ανάγκες ε, γίνονται ακόμα πιο έντονες στους νέους. Και ε, τα κοινωνικά παντοπολία ε, είναι κάτι που τους αφορά ιδιαιτέρως οι ανάγκες τους ε, είναι όλο και πιο οξυμένες. Εξαιρετική ιδέα λοιπόν να έχουμε στατιστικές αναφύλλο, ζητώ όμως να έχουμε ε, και στατιστικές αναπληθυσμιακή ομάδα, αναηλικία. Τρίτον, ή τέταρτον δεν θυμάμαι. Η κυρία Εντίτ Μπάουερ είπε ότι αυτό το ταμείο είναι εξαιρετικά ελληματικό, ανεπαρκές και ε, βεβαίως συμφωνώ απολύτως. και η κυρία Κώστα το είπε πρόλίγου. Για να παραμείνουμε στα προηγούμενα επίπεδα και να έχουμε σκιαγραφίσει συγκεκριμένη ε, περίμετρο ε, των δράσεών μας αλλά και των χωρών οι οποίες θα εμπλακούν, θα έπρεπε να είχαμε διατηρήσει 3,5 δις και αυτή τη στιγμή είμαστε στα 2,5 δις από ή και ένα Βλέπετε λοιπόν την περικοπή την τεράστια. Και τώρα, όσο και αν είμαστε μέλη στις διαφόρες επιτροπές, τόσο περισσότερο πρέπει εκεί να ε, τονίζουμε το γεγονός ότι τα γεωργικά πλεονάσματα, τα οποία συνεχώς συνεχίζουν να υφίστανται, θα πρέπει ρητά και πολύ συγκεκριμένα να αναδιοχετεύονται προς τους πιο ενδεείς συνανθρώπους μας, ούτω ώστε να αντισταθμίσουμε εν μέρη, πάρα πολύ εν μέρη, την ριζική ε, περικοπή αυτού του ταμείου. Και τέλος, σίγουρα θα συμφωνείτε, ως προς το εξής. Ως εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, για τα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, ε, συνεχώς μου ζητούν, για να μην πω τίποτα χειρότερο, να ε, τοποθετηθούμε αναλόγως ε, με τα νέα στοιχεία. Και νομίζω ότι η Επιτροπή μπορεί να, ε, να το διαψεύσει αυτό. Λοιπόν, παίρνουμε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για να δώσουμε στους φτωχούς. Δηλαδή παίρνουμε από τη μία τσέπη των φτωχών για να τα βάλουμε στην άλλη δεν αυξάνεται αλλά μειώνεται. Αυτό μας φέρνει όλους σε μια πολύ δυσχερή θέση. Οι αρχικοί κρατών και κυβερνήσεων μετά τη σύνοδο βγήκαν και είπαν ότι εμείς σώσαμε το Ταμείο Ενίσχυσης των πιο ενδεών. Ναι, το έκαναν, αλλά με περικοπές στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, του οποίου ο μέγιστος στόχος είναι η κοινωνική ενσωμάτωση μέσα από την επαγγελματική ένταξη. Ουσιαστικά, στερήσαμε από τους φτωχούς τα φτωχά του σημάτια για να τους θρέψουμε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Κορνέλισεν, για την σκληρή της δουλειά. Εν μέρη συμφωνώ με τη γνωμοδότηση. Το ζήτημα είναι περίπλοκο. Πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη στους απόρους, ιδιαίτερα τις γυναίκες και τα παιδιά που βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Ο καθένας χρειάζεται βασικό ρουχισμό και τροφή και σε αυτό το σημείο εδώ μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει μέσω του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους. Σημαντικό είναι να μην παρέχει μόνο άμεση βοήθεια η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και να στηρίξει τις τοπικές συνδέσεις ανάμεσα στους ε, παραγωγούς τροφίμων και τους οργανισμούς αυτούς. Οι γυναίκες επλήγησαν περισσότερο από όλους από την φτώχεια. Γι' αυτό και εκείνες είναι αυτές που θα βοηθήσει περισσότερο το ταμείο αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, ολοκληρώσαμε λοιπόν τη συζήτηση για το σημείο αυτό. Κύριε Κορνέλισεν, έχετε το λόγο ή... Όχι, η κυρία Ζούμπερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ως προς το ταμείο αυτό, η συζήτηση αυτή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της και την ανάλυση του πώς εξελίσσεται η φτώχεια σήμερα στην Ευρώπη. Παρόλο που είναι ένα φαινόμενο που έχει λάβει καινούριε διαστάσεις. Οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης έχουν παρόμοια προβλήματα πλέον. Όμως, τα ποσοστά φτώχειας που βλέπουμε σήμερα σε πολλές χώρες, ιδίως στις περιφέρειες της Ευρώπης, και κυρίως όσες έχουν, ε, βρίσκονται στο καθεστώς προγράμματος της Τρόικας, αυτά είναι διαφορετικά στοιχεία από ότι θα μας απασχολούσε σήμερα και θα μας απασχολήσει την επόμενη πτέτεια από το 2014 στο 2020. Σήμερα μιλάμε για αύξηση τη φτώχεια σε οικογένειε που ουδέποτε είχαν αντιμετωπίσει αυτό το ε, ενδεχόμενο, ουδέποτε είχαν φανταστεί ότι μπορεί να ζήσουν σε συνθήκε φτώχεια. Αυτό είναι κάτι τελείω διαφορετικό. Μιλάμε για οικογένειε που γνώρισαν, δεν μιλάμε για οικογένειε που γνώρισαν την ανεργία, τη διαρθρωτική, την μόνιμη εδώ και χρόνια, αλλά ανθρώπου που βρέθηκαν ξαφνικά στη φτώχεια γιατί βρέθηκαν ξαφνικά άνεργοι. Ή ένα από τα μέλη τη οικογένεια ε, βρέθηκαν άνεργα, ή δουλεύουν μεν, αλλά δουλεύουν σε συνθήκε φτώχεια. Δηλαδή με μισθού που είναι τόσο χαμηλοί, οι οποίοι πραγματικά του φέρνουν κάτω από το κατόφλι τη φτώχεια. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που δεν μπορούμε. Ε, είναι πολύ διαφορετική φτώχεια σήμερα. Τα άτομα που έχουν επενδύσει σε ένα στεγαστικό δάνειο λόγω χάρη όλη του τη ζωή, ξαφνικά βρίσκονται να μην μπορούν να πληρώσουν στην τράπεζα και να βρίσκονται στο δρόμο. Ε, κάτι άλλο που μα απασχολεί και τώρα στην Πορτογαλία είναι η παιδική φτώχεια. Ο αριθμό των παιδιών που πάνε σε σχολείο και έχουν ένα μόνο από το σχολείο, αυτό είναι κάτι που είναι πραγματικά δραματικό πλέον. Η συζήτηση λοιπόν για το ταμείο αυτό θα πρέπει να γίνει με όρους πολύ σοβαρούς. Εάν δεν ε, δούμε όμως τη διάσταση ότι η φτώχεια και απλώς δεν μειώνεται, αλλά αλλάζει και μορφή σε σχέση με το φαινόμενο όπως το γνωρίζαμε ως τώρα, δεν θα πετύχουμε τίποτα. Κανείς δεν θα καταλάβει ούτε η κοινή γνώμη, ούτε κανένα πολίτη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υποθέτει στόχου ε, για τι διαφορετικέ χώρε, μειώνοντα όμω του μισθού, μειώνοντα τι δημόσιε επενδύσει, μειώνοντα την κοινωνική προστασία. Και όταν έχει μια δυνατότητα να αναχαιτήσει κάποιε από τι διμερεί επιπτώσει αυτών των αρνητικών πολιτικών, ε, δεν τηρεί τις ίδιες αξίες ε, για την πραγματική καταπολέμηση της φτώχειας. Νομίζω λοιπόν ότι η γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου θα έπρεπε να αναφέρεται στο εξή. Να διατηρήσει ή τουλάχιστον να επιτρέψει τα κονδύλια που ήδη προβλέπονταν ανά έτος, ή να υπάρξει διαφοροποίηση των δράσεων του Ταμείου. διότι θα πρέπει να δικαιολογείται η αύξηση που ζητούμε για το Ταμείο. Ιδάλω δεν θα εξασφαλίζεται ούτε κάνει η βοήθεια. Νομίζω ότι το Ευρωκοινοβούλιο λοιπόν θα πρέπει να έχει μια σαφή τοποθέτηση στι διάφορε επιτροπέ που ασχολούνται με την έκθεση αυτή. Διότι τουλάχιστον θα ήταν μια εξελαχή στον τοποθέτηση που θα μπορούσε να αποδείξει ότι κάπως εδώ προστατεύουμε, συμφιλιώνουμε με τις απόψεις μας την προστασία των βασικών δικαιωμάτων για ανθρώπους που βρέθηκαν σε μια κατάσταση την οποία ουδέποτε είχαν προγραμματίσει. Μιλάμε για διαφορές σε σχέση με τη διαδοτική ανεργία που, τόσο, που μέχρι τώρα γνωρίζαμε. Ευχαριστώ. Και τώρα για να κλείσει η συγγήτρια, κυρία Κορνέλισον. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας και τις προτάσεις σας. Να σχολιάσω αυ... αυτό... αυτή την κατανομή των πόρων. Πολλοί είπαν ότι είναι γελία αυτή η μείωση των κονδυλίων του Ταμείου να αυξάνεται η φτώχεια και αυτό είναι αλήθεια. Δυστυχώ όμω δεν μπορούμε να κάνουμε σε αυτήν εδώ την Επιτροπή πάρα πολλά. Ούτε η Επιτροπή απασχόληση μπορεί να κάνει πολλά, η οποία είναι και η Επιτροπή επί της ουσίας, διότι αυτό θα αποφασιστεί στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων. Αυτό που πιστεύω είναι ότι τώρα δεν έχουμε 2,5 δισεκατομμύρια, αλλά 2,1 δισεκατομμύρια ως κονδύλια. Ελπίζω να αυξηθεί το ποσό αυτό και θα πρέπει να πάρουμε αυτά που έχουμε στην παρούσα φάση. Αυτό που προσπάθησα να κάνω με αυτή τη γνωμοδότηση είναι να κατευθύνω τα κονδύλια στις χώρες οι οποίες τα χρειάζονται περισσότερο. Εάν φυσικά υπάρχει ανάγκη σε όλες τις χώρες και τα κονδύλια είναι επαρκή, τότε ναι, να διαμοιραστούν σε όλες. Αλλά πρώτο στο μέλημά μας είναι τα κονδύλια αυτά να πάνε εκεί που χρειάζονται περισσότερο. Η κυρία Ζούπερ μόλις μας έδωσε μία ολοζώντανη εικόνα του πόσο άσχημη είναι η κατάσταση σε ορισμένες χώρες. Ε, επίσης υπάρχουν πάρα πολλές ε, χώρες στις οποίες έχει αυξηθεί ο αριθμός των εξαρτημένων ατόμων και εκεί θα έπρεπε να πάνε τα κονδύλια αυτά. Τώρα, όσον αφορά την τροπολογία 30 που ανέφερε και η κυρία Μπάουερ, να πω ότι εκεί προσπάθησα να κάνω έναν διαχωρισμό. Δηλαδή, οι πλουσιότερες χώρες πρέπει να παρέχουν οι ίδιες κονδύλια για τους απόρους και τα κονδύλια του Ταμείου να πάνε στις ε, φτωχότερες χώρες, εκεί που χρειάζονται περισσότερο. Στην τροπολογία 30 αναφέρεται στο τέλος ή το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Δεν θα έπρεπε να το λέει, να διορθώσω, θα έπρεπε να λέει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής. Οι χώρες συνοχής λοιπόν είναι αυτές που θα έπρεπε να πάρουν περισσότερη συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ οι χώρες που δεν ανήκουν ούτε στι χώρε συνοχή, ούτε στις χώρες ε, σταθερότητας θα πρέπει να συνεισφέρουν, να πληρώσουν περισσότερα έτσι ώστε τα χρήματα αυτά να πάνε στις χώρες που τα χρειάζονται. Τώρα, συμφωνώ με όλους όσους ε, είπαν ότι... ότι η συγκέντρωση, η επικέντρωση μάλλον στα τρόφιμα δεν θα λύσει το πρόβλημα και υπάρχει ανάγκη και σε άλλους τομείς εκτός από τα τρόφιμα και εκτό από το να διευρύνουμε το ταμείο, μπορούμε να κάνουμε και άλλε δραστηριότητε. Για παράδειγμα, να δώσουμε στου διάφορου φορεί περισσότερε επιλογέ στο πώ θα χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια. Τώρα, το σχολείο τη κυρία Μωράν Σαχτιέ για το εάν το ταμείο είναι περισσότερο για γυναίκε. Δεν το εννοώ έτσι ακριβώ. Δεν εννοώ ότι θα έπρεπε να είναι ταμείο για τις γυναίκες, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή. Η πικρή αλήθεια είναι αυτή. Δυστυχώς οι περισσότεροι άποροι είναι γυναίκες. Και αυτό ως Επιτροπή μας δίνει δικαίωμα να μιλήσουμε και να επηρεάσουμε τις συζητήσεις και την εξέλιξη αυτού του ταμείου. Επίσης, να κοιτάξουμε και τα υπόλοιπα σχόλια. Καλό θα είναι να έχουμε μια συνάντηση των σκιωδών εισηγητών, διότι έχουμε πάρα πολλές επιλογές, υπάρχουν πολύ διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης. Είμαι σε, στην επαφή με την κυρία Κοστέλο, η οποία είναι και η κύρια εισηγήτρια της Επιτροπής Απασχόλησης και πιστεύω ότι πολλές συζητήσεις εντός και εκτός Επιτροπής πρέπει να συνεχιστούν έτσι ώστε το Ταμείο αυτό να συσταθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να κάνουμε την ευέλτιστη δυνατή χρήση των πόρων που διαθέτουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να σας δώσω το χρονοδιάγραμμα για το θέμα αυτό. Προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών 25 Φεβρουαρίου στις 5 το απόγευμα. Η Επιτροπή θα ψηφίσει στις 20 Μαρτίου και η Επιτροπή Απασχόλησης 23 Απριλίου. Και τώρα να προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, εκπαιδευτική και επαγγελματική κινητικότητα των γυναικών στην Ευρώπη. Να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, την κυρία Ραντσούλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τους συναδέλφους, όλες τις συναδέλφους που συνεισέφεραν για την σύνταξη αυτής της ωραίας κατά την απόψή μου έκθεσης. 103 τροπολογίες που αφορούν αιτιολογικές σκέψεις και άρθρα. Θα ξεκινήσω από τις αιτιολογικές σκέψεις. Πολλές ήταν οι προτάσεις των συναδέλφων που επαναλαμβάνουν και υπογραμμίζουν έννοιες που ήδη περιλαμβάνονται στο διατακτικό του αρχικού κειμένου. Έμφαση δίνεται στην ελευθερία των πολιτών, των Ευρωπαίων πολιτών, να διαμένουν και να εργάζονται ελεύθερα σε όλη την Ευρώπη, κάτι που προφανώς το παρέχει η επαγγελματική κινητικότητα, ενισχύοντας το συνέστημα του ανήκειν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. στις συνεισφορές αυτές, όπως και στο αρχικό κείμενο, υπογραμμίζεται η διαφορά μισθών στους μισθούς, η δυσκολία συμφιλίωσης επαγγελματικού και γενιακού βίου και η έλλειψη, το, η των ε, βρεφονιπιακών σταθμών Κάτι που δυσκολεύει πολλέ φορέ την επίτευξη ακριβώ τη συμφιλίωση που μόλι ανέφερα. Σε ό,τι αφορά τα άρθρα, θα είμαι πιο συγκεκριμένη. Οι τροπολογίε από την 23 ω την 31 προτείνουν την... στην συμπερίληψη του άρθρου 1 την αναφορά στο ότι η γυναίκα πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο των ευρωπαϊκών πολιτικών σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, την απασχόληση και τη μετανάστευση. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέροντα εφαλτήρια για να σκεφτούμε και να στα συμπεριλάβουμε και όλα σε μια συμβαστική τροπολογία στις τροπολογίες 32 ως 41 αναφέρονται αυτές στο άρθρο 2 του αρχικού κειμένου ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων των γυναικών στο πλαίσιο της επαγγελματική κινητικότητας διασφαλίζοντας και τα δικαιώματα στη σύνταξη οδότηση ανταλλαγή καλών πρακτικών επίσης ε, και προστασία της ισότητας των φύλων. Νομίζω και αυτά μπορούν να συμπεριληφθούν σε μια συμβαστική τροπολογία. Τροπολογίες από 42 έως 47. Άρθρο 3. Δυσκολία των γυναικών στην εξέβρεση εργασίας σε άλλη χώρα. Τροπολογίες 48-53. Εδώ επιμένουν στο άρθρο 4 για την παροχή θέσεων με χαμηλούς μισθούς, υποβιβαστικές ε, πολλές φορές, στις γυναίκες κατά κύριο λόγο. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να εκφράσω την αντίρρησή μου. Κυρίως ως προς την τροπολογία 48 της συναδέλφου Τσέσκοβα η οποία ζητά την διαγραφή ολόκληρου του άρθρου. Εδώ την έχω. Και αυτό γιατί δεν πιστεύω ότι η κατάργηση ενός εδαφείου, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, προσφέρει κάτι παραπάνω στην έκθεση. Και επειδή ακριβώς δεν μου φαίνεται και σωστό αυτό. Στην ουσία το συζητάμε από καιρό ε, το θέμα αυτό, την διαφορά μισθών μεταξύ ανδρών και γυναικών καλό θα ήταν να παραμείνει το εδάφιο. Επίσης έχω πολλού συνδυασμού για την τροπολογία 50 της συναδέλφου τριβέτη. Εδώ καλούνται τα κράτη-μέλη να εξεύρουν λύσεις για να προλαβούν να αντισταθμίσουν τι επιπτώσει που προκύπτουν από την επαγγελματική κινητικότητα σε αυτά τα κράτη-μέλη σε συγκεκριμένου τομεί όπω την κινητικότητα των ε, ιατρικών ε, εργαζομένων Κάτι που δεν προστατεύεται παρκώς και κυρίως αφορά γυναίκες και μπορεί να αποτελεί και παράβαση του δικαίου της χώρας προέλευσης. Καμία, κανένας επαγγελματικός κλάδος δεν θα έχει δικαίωμα στην κινητικότητα εάν η επαγγελματική κινητικότητα δεν προσέφερε συγκεκριμένα ωφέλη σε επαγγελματικού κλάδου, σε πολλού επαγγελματικού κλάδου. Το ότι από καιρό, ε, καιρόν λείπει συγκεκριμένους ε, αριθμός γυναικών στη συγκεκριμένη περίπτωση από κάποιους κλάδους, αυτό είναι κάτι προσωρινό. η αρχή αυτή δεν είναι κάτι που μπορεί να ισχύει για όλους τους επαγγελματικού κλάδους. Μπορεί να συμβαίνει στις ε, ιατρικές υπευθύνου, αλλά όχι για όλους του επαγγελματικού κλάδους. Από την 50 65, την τροπολογία 50 65, μιλάμε για την προστασία συγκεκριμένων δικαιωμάτων των γυναικών για την αγορά εργασία. Εδώ πρέπει να πω για την τροπολογία 60 και επειδή μιλά για το ποσοστό της εργασίας σε μερικό χρόνο και την διαφορετική συμμετοχή στην εργασία αυτή ανδρών και γυναικών, αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το δούμε. Οι τροπολογίε 61, 62, 63 που αφορούν το άρθρο 6 για την καταπολέμηση της διακριτική μεταχείριση, έμεση ή άμεσης, και αυτό, όπως προηγουμένω έλεγα, είναι κάτι που ζητά κατάργηση μέρους ενός άρθρου, ενό εδαφείου. Όπως είπα και προηγουμένω δεν είμαι υπέρ τη ε, απάλληψης ολόκληρων άρθρων. σε ό,τι αφορά το άρθρο 8 της τροπολογίας 65 και 70 δεν νομίζω ότι οι συλλογικές συμβάσεις είναι χρήσιμο εργαλείο για να αντισταθμιστούν οι αποκλήσει οι μισθολογικές. Αυτό για τη συνάδελφο Ζούμπερ. Ούτε θα πρέπει να προβλεφθεί υποχρέωση για τους εργοδότες να υποβάλουν στατιστικά στοιχεία για την διαφορά τη μισθολογική όπως κατανέμεται μεταξύ των φύλων. Ακριβώς πάλι η τροπολογία 70. Μία συμπαρατήρηση και για την τροπολογία 80, για το άρθρο 11 τη συναδρέφου Γκριμπόφκα. Εδώ νομίζω ότι πρέπει να υπήρξε ένα μεταφραστικό πρόβλημα ή έστω ένα πρόβλημα στην έκφραση στα Ιταλικά, όπου γίνεται λόγος για την αναγνώριση διαμονής στο εξωτερικό προκειμένου οι συνταξιδοτικέ να συνυπολογιστούν στο μέλο προέλευση. Δεν ξέρω, ίσως θα μπορούσαμε να βρούμε μια άλλη ορολογία, πιο εύστοχη, αλλά δεν αναφερόμαστε αναγκαστικά με τη διαμονή στο εξωτερικό σε διακοπές, ας πούμε, αλλά σε μια περίοδο άσκησης, ένα στάζ στο εξωτερικό εργασιακό. Τώρα για κάποιε τροπολογίε που. Αναφέρομαι μάλλον κυρίω στι τροπολογίε οι οποίε μου δημιουργούν κάποιε δυσκολίε. Τι άλλε προφανώ θα χρειαστεί να σταθώ. Για την τροπολογία 113 και καταλαβαίνω ότι αυτή είναι προσωπική μου άποψη και εδώ ίσως να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Δεν έχω όμως πρόβλημα να αναφέρω τι πιστεύω και στην Επιτροπή μας. Το άρθρο 13 μάλλον. Ε, τροπολογίες από την 93 έως την 97, ιδίως η 95 της συναδέλφου Κλειβέτη, δεν μου φαίνονται να αναφέρονται σωστά στο εξή, που το λέω εδώ και τέσσερα χρόνια και σε άλλες επιτροπές για παρόμοιες εκθέσεις. Εδώ αναφέρεται κάτι που το βρίσκω αναρθόδοξο. Δεν μου φαίνεται δίκαιο να αναφέρουμε. Δεν το βρίσκω σωστό μάλλον να αναφέρουμε την εθνική προέλευση των ε, Ρώμα. Ή θα αναφέρονται όλε οι μειονότητε ή θα κάνουμε μια εξαίρεση. Εάν θέλουμε να αναφερόμαστε στην εθνοτική μειονότητα των Ρωμά, να σας πω την αναφέρει και η τροπολογία. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και να αναγνωριστεί αυτή η ανάγκη στη στήριξη της κινητικότητας των γυναικών άνω των 45 ετών οι οποίε είναι εκτεθειμένες περισσότερο από άλλε στο να αποδεχτούν επισφαλεί θέσει εργασία. Ωστότε, ωστό εδώ θα ήταν καλό το κείμενο, αλλά ολοκληρώνει λέγοντα να εξεύρουμε συγκεκριμένε λύσει για να επιλύσουμε τα προβλήματα των γυναικών Ρώμα. Νομίζω ότι εδώ δείχνουμε ιδιαίτερη διακριτική μεταχείριση, τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου προσωπική σκοπιά. Δεν ξέρω αν είναι μόνο προσωπική άποψη, είμαι μονομένη. Θα το δούμε. Νομίζω τα κάλυψα όλα. Να ευχαριστήσω και πάλι τις συναδέλφους και τους συναδέλφους που συμμετείχαν στην επεξεργασία αυτού του κειμένου και ελπίζω πολύ σύντομα να μπορώ να σας στείλω προτάσεις για συμβαστικές τροπολογίες. Ευχαριστούμε. Και τώρα να δούμε τρεις ε, ομιλητέ στον κατάλογο των αγορητών. Απλώς να σας πω ότι δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Να σας ευχαριστήσω κυρία Ροντζούλη. Είναι μια πολύ καλή βάση αυτή που μας παρουσιάσετε για την έκθεση αυτή. Αυτές οι δυσκολίες αφορούν όλο και περισσότερους ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσωπικό συμφωνώ και με τις 103 τροπολογίες για πολλούς και διάφορους λόγους. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη στην παράθεση των λόγων. Θα πω τα μισά από αυτά που θα ήθελα να, είχα, να πω. Η τροπολογία για την προστιθέμενη αξία της κινητικότητας είναι πολύ σημαντικό για τους Ευρωπαίους πολίτες. Ειδικά που φέτος είναι η χρονιά των Ευρωπαίων πολιτών. Οι τροπολογίες ε, μεταξύ των, που έχουν να κάνουν με τα διάφορα κοινωνικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ σημαντικό αυτό. Δεν εκπρόσωπο βέβαια την κυρία Ζαμπόρσκα, αλλά η τροπολογία της είναι πολύ σωστή. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε κάτι τέτοιο και να προβληματιστούμε. Μισθολογική ανισότητα αναφύλλω, συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και εργασιακής ζωής. Πολύ σημαντικά αυτά. Ανάγκη για περισσότερες και μεγαλύτερες γλωσσικές δεξιότητες. Όλα αυτά τα στηρίζουμε, είναι πολύ καλά. Τώρα ως προς τις δικές μου τροπολογίες, αποδοχή διπλωμάτων. Πολύ σημαντικό συζητείται πολύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα πρέπει να λυθεί αυτό το θέμα περιπτώσει και να υπάρχει σε κάθε έκθεσή μας αυτό το αίτημα και η ύπαρξη περισσότερων γυναικών στις επιτελικές θέσεις, στις θέσεις όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις και αυτό είναι υποσυζήτηση αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολύ σημαντικό. Κινητικότητα για εκπαιδευτικούς λόγους των γυναικών και ειδικότερα ε, κινητικότητα στην ανώτερη εκπαίδευση. Μιλώ για τις καθηγήτριες κυρίως πανεπιστημίου, που δεν είναι και τόσο πολλές. Υποεκπροσωπούνται οι γυναίκες γενικότερα και υποεκπροσωπούνται και στις ανώτερες εκπαιδευτικές βαθμίδες. Το πρόγραμμα εγγύησης των, στους νέους, το Youth Guarantee Scheme, είναι πολύ σημαντικό ε, οι γυναίκες να εκπροσωπηθούν εκεί. Άνω του 50% των πτυχιούχων αυτή τη στιγμή είναι γυναίκες και θα πρέπει να διευκολύνεται η πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας. Και μέσω αυτού του προγράμματος για τους νέους ε, μπορούμε να ενισχύσουμε την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας και εθελούσιες εθελοντικές δραστηριότητες για ανταλλαγή βιωμάτων, εμπειριών μεταξύ διαφόρων ε, πληθυσμιακών ομάδων για να γνωρίζουν καλύτερα οι άνθρωποι τι μπορούν να περιμένουν από την κινητικότητα και να ενισχυθεί αυτή που είναι μία από τις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Επόμενη ομιλήτρια η κυρία Κλεβέτη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ την εισηγήτρια η οποία έκανε εμβρηθή ανάλυση των τροπολογιών, κάτι το οποίο είναι πολύ καλό. Να πω καταρχάς ότι επιθυμώ να συνεργαστώ με την εισηγήτρια για να εξηγήσουμε ακόμα περισσότερο, να διευκρινίσουμε μάλλον καλύτερα ορισμένα προβλήματα. Εν συντομία λοιπόν θα πω τα εξή. Είναι αληθές ότι είμαι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά εκπροσωπώ και τη χώρα μου. Προφανώς όλοι το ίδιο κάνουμε. Αυτό το οποίο με ενδιαφέρει είναι η ύπαρξη δύο κατηγοριών τροπολογιών, οι οποίες καλό θα είναι να συζητηθούν περισσότερο. Δηλαδή, τροπολογίες που αφορούν στους γιατρούς. Στη χώρα μου, για παράδειγμα, η πλειονότητα των γιατρών είναι γυναίκες και πολύ κινητικές ε, στο επαγγελματικό πεδίο, κάτι το οποίο είναι καλό. Δεν είναι πρόθεσή μου να πω ότι πρέπει να ε, μην επιτρέπουμε στις Ρουμάνες γιατρούς να εγκαταλείπουν τη χώρα τους ή να κινούνται γενικότερα, αλλά από την άλλη δεν θα πρέπει να εγκαταλείψουμε και τους ασθενείς στη χώρα μου. Θα, καλό θα είναι λοιπόν σε κάθε έκθεση να προσπαθούμε να ε, μεριμνούμε έτσι ώστε να βρίσκονται λύσεις γενικότερα. Αυτό είναι μια λύση που που προτείνω στην τροπολογία μου και γι' αυτό την υπέβαλα, την τροπολογία αυτή. Ως προς τους πληθυσμούς Ρωμά, συμφωνώ, πρέπει να έχουμε ξεχωριστή έκθεση για να επιλύσουμε όλα τα προβλήματα των γυναικών που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Αλλά όπως και να έχει το πράγμα, το πρόβλημα παραμένει για τη δική μου χώρα και γι' αυτό δεν διστάζω να το προσεγγίσω το πρόβλημα αυτό κάθε φορά που προκύπτει σε οποιαδήποτε έκθεση. Τα λέω αυτά για να εξηγήσω τη στάση μου στην εισηγήτρια, την οποία ευχαριστώ θερμά διότι ανέλησε τα προβλήματα αυτά τα οποία αφορούν δυστυχώς ε, ειδικά τη δική μου χώρα. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος και εγώ σας ευχαριστώ η κυρία Σούπερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι κατά την άποψή μου η έκθεση αυτή είναι πολύ σημαντική και το ζήτημα το οποίο μας απασχολεί είναι εξίσου σημαντικό. Το λέω αυτό διότι σήμερα η μετανάστευση παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις όχι μόνο διότι αυτό είναι επιθυμία των ατόμων, επιθυμούν να πάνε να εγκατασταθούν αλλού, αλλά μερικές φορές και πολύ συχνά μάλιστα υποχρεούνται, αναγκάζονται να εγκατασταθούν αλλού για να βρουν δουλειά και πρέπει να εγκαταλείψουν την οικογένειά τους, τις ρίζες τους και αυτό για να βρουν δουλειά. Θα πρέπει λοιπόν οι χώρες υποδοχής να τους υποδέχονται με τρόπο αξιοπρεπή, με κατά πώς τους ταιριάζει. Ως προς την οικογενειακή επανένωση λοιπόν. Είναι κάτι το πολύ σημαντικό για τις γυναίκες. Είναι ένα δικαίωμα προφανώς η οικογένεια να μπορέσει να βρει τη γυναίκα που μεσταναστεύει. Αυτό είναι προφανές. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να δημιουργήσουμε και τις κατάλληλες συνθήκες έτσι ώστε και ο σύζυγος να βρει δουλειά θα πρέπει να υπάρχει ένα δημόσιο δίκτυο πρόσβασης για τα παιδιά, να έχουν τα παιδιά πρόσβαση ε, στις υποδομές, στους βρεφονιπιακούς ε, σταθμούς, νηπιαγωγείο, σχολείο και του καθεξής. Αυτά ήθελα να προτείνω για αυτή την έκθεση και θα ήθελα να υπογραμμίσω το πόσο σημασία έχει η προώθηση των συλλογικών συμβάσεων. Μιλήσαμε για τις μισθολογικές ανισότητες και την ανάγκη εξάλληψής τους. Και θα πρέπει να βρούμε μέτρα εύστοχα για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Τώρα για τις αποχρεώσεις ε, για τους εργοδότες, εγώ να προσθέσω εδώ ότι υπάρχουν ε, εργαζόμενοι οι οποίοι εργάζονται με συμβάσεις, οι, οποίοι δεν, ε, οι οποίες δεν εφαρμόζονται με τέτοια κριτήρια για όλες τις επαγγελματικέ ομάδες ή για όλους τους εργαζομένους. Θα πρέπει οι συμβάσεις να είναι και διαφανέστερες και να είναι δημόσιες, ε, να είναι δημόσια τα κριτήρια και οι όροι πρόσληψης. Κάτι που να το γνωρίζουν όλοι οι εργαζόμενοι και υποψήφοι. Αυτό είναι σημαντικό και για τις γυναίκες και είναι πολύ πιο εύκολο χωρίς να υπάρχει διαφάνεια να υπάρξει και διακριτική μεταχείριση. Προφανώς αν δεν γνωρίζουν ποιοι είναι οι μισθοί που προσφέρονται στους υπόλοιπους εργαζομένου, μπορεί να υπάρξει διακριτική μεταχείριση. Θα πρέπει λοιπόν να καταπολεμηθεί η μισθολογική ανισότητα και να στηρίξουμε αυτό το μέσο. Ένα μέσο που να προστατεύσει και τις γυναίκες κατά των ε, διακριτικών συμπεριφορών. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σόρτια έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, πολύ γρήγορα. Καταρχάς να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εργασία της, η οποία και εντατική ήταν και πολύ ακριβής η παρουσίαση των συνεισφορών των διαφορών πολιτικών ομάδων μέσω των τροπολογιών. Να επιμείνω σε ένα σημείο. Όλοι βεβαίως θέλουμε να αναλάβουμε δράση προκειμένου να στηρίξουμε την επαγγελματική κινητικότητα των γυναικών στην Ευρώπη και να μπορέσουν και εκείνε όπω όλοι οι εργαζόμενοι να συμμετάσχουν σε αυτήν την κίνηση, την ε, μαζική κίνηση που υπάρχει μέσα στα κράτη-μέλη. Αλλά εδώ θα πρέπει να δούμε και την ανάγκη οι σταδιοδρομίε των γυναικών να συνεχίσουν να υποστηρίζονται. Και είναι πολύ απαιτητικέ πολλές φορές, διότι η κινητικότητα μεταξύ χωρών επιφέρει μια τελμάτωση κάποιες φορές και πολλές φορές και οπισθοδρόμηση στη σταδιοδρομία των γυναικών. Πολλοί από εσά αναφερθήκατε στα προβλήματα μισθολογική ανισότητας. Το πρώτο πρόβλημα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι ανισότητε στην επαγγελματική ανέλυξη. Οι γυναίκες έχουν τα ίδια εκπαιδευτικά προσόντα με τους άντρες. Ε, οι νέε γυναίκες είναι εξίσου ικανέ με τα νέα με τους νεαρούς άντρες, όμως η ανισότητα επαγγελματικών ευκαιριών που προσφέρονται είναι απαράδεκτες σε σχέση με το, με το πόσο εκπαιδευμένοι είναι οι πολίτες μας. Εδώ λοιπόν θα πρέπει με τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί και στην προσοχή που πρέπει να δοθεί στην ε, ισότητα των ε, ευκαιριών σταδιοδρομίας είναι κάτι που όλοι θα πρέπει να στηρίξουμε. Ευχαριστώ. Κάποιος από την Επιτροπή που θα ήθελε το λόγο για αυτό το σημείο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον Πρόεδρο, την εισηγήτρια και τα αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου για την, τον συντονισμό της έκθεσης αυτής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσορίζει την πρωτοβουλία αυτή και το περιεχόμενο της ε, έκθεσης και τις ατροπολογίες οι οποίες, δίνουν τροφή για συζήτηση. Η έκθεση αυτή εστιάζει ιδιαίτερα σε ζητήματα τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί πρωτής της σημασίας στην πολιτική της, δηλαδή την διαβίου μάθηση, για παράδειγμα, την παιδική μέρημνα, την αντιμετώπιση της μισθολογικής ανισότητας, της εγγύησης για τους νέους. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την τελευταία περίοδό της. Ε, τώρα θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια όσον αφορά την απασχόληση και την κινητικότητα και ο συνάδελφός μου θα σας ε, σχολιάσει τις απόψεις ε, που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση. Να τονίσω ότι η έκθεση για μας πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Για μας είναι για μας η ενεργοποίηση των γυναικών είναι πολύ σημαντική για το στόχο της πληθυσμιακής ομάδας 64. Τώρα, κοιτάζοντας τα στατιστικά στοιχεία, βλέπουμε ότι οι άνδρες ε, κοντεύουν να φτάσουν αυτό το στόχο του 75% των... σε θέσεις εργασίας. Και η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας είναι θεμελιώδης έτσι ώστε να φτάσουμε το στόχο του συνολικού 75% στην αγορά εργασίας. Σε ορισμένες χώρες πρέπει να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών, διότι υπάρχει πολύ χαμηλή συμμετοχή τους στην αγορά εργασία. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνουμε το θέμα πολύ σοβαρά υπόψη και θα λάβουμε υπόψη και τις ε, τροπολογίες και την ίδια την έκθεση. Πολλά από αυτά τα ζητήματα αφορούν, όπως είπα, τις, ε, την επαιδική μέρημνα, την μισθολογική ανισότητα, τα δικαιώματα στις συντάξεις και την διαβίου μάθηση και κατάρτιση, αλλά και την κινητικότητα και την επαγγελματική κινητικότητα. Αυτό είναι μέρος της ε, πολιτικής μας για την διασυνοριακή και κινητικότητα. Τώρα, θα ήθελα να σας παραπέμψω στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και τις συστάσεις αναχώρα που έχουν ήδη εκδοθεί το 2012 για ορισμένα κράτη-μέλη Και να αναφερθώ ότι η Αυστρία, η Γερμανία, η Ουγγαρία, η Τσεχία, η Πολωνία και η Σλοβακία και το Ηνωμένο Βασίλειο μεταξύ άλλων έχουν λάβει συστάσεις τέτοιες Επίσης, στην Γερμανία και στις 100 χώρες έχουν γίνει ιδιαίτερες συστάσεις για την απασχολησιμότητα καθώς και έχουν γίνει συστάσει στην Αυστρία για τη μισθολογική ανισότητα ανδρών και γυναικών. Φέτος θα ασχοληθούμε με την κινητικότητα και τη δυσκολία στην ε, επαγγελματική κινητικότητα και την ε, διαβίου μάθηση και τις διάφορες απόψεις της. Τώρα, όσον αφορά την γεωγραφική κινητικότητα, να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Νοέμβριο εξέδωσε μία απόφαση, μια πλατφόρμα, δημιούργησε μια πλατφόρμα στην οποία εκλήθησαν τα κράτη-μέλη να την χρησιμοποιήσουν να τις χρησιμοποιήσουν κυρίως οι γυναίκες και να τη χρησιμοποιήσουν επίσης για να αντιμετωπιστεί η ανεργία. Η ανεργία η οποία πλήττει κυρίως τις γυναίκες όπως έχουμε πει. Κλείνοντας, θα αναφερθώ στις ε, συντάξεις και τη δυνατότητα μεταφοράς των συντάξεων. Η δυνατότητα αυτή έχει δύο διαστάσεις. Η μία διάσταση έχει να κάνει με τον κατακαιρματισμό της αγοράς εργασίας και να σας πω ότι μόνο ένας στους δέκα άνδρες εργάζεται σε η απασχόληση ή εθελοντικά ή προσωρινά. Και πολλές από τις διακρίσεις στον τομέα των συντάξεων σχετίζονται με τα δικαιώματα που έχουν προκύψει από αυτόν τον κατακαιρματισμό της αγοράς εργασίας. Αρχίσαμε να εργαζόμαστε πάνω σε αυτό κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας και τώρα η Ιρλανδική Προεδρία έχει προγραμματίσει αρκετές συνεδριάσεις για το, τη μεταφορά των συντάξεων. Τώρα θα δώσω το λόγο στον συνάδελφό μου, στην συνάδελφό μου μάλλον. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Ως εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης να ευχαριστήσω την κυρία Ροντσούλη για την έκθεση αυτή. Να πω ότι και εμεί καλωσορίζουμε την έμφαση που δίνει η έκθεση στον κανόνα εκπαίδευση και παιδεία να παρέχονται στι γυναίκε προκειμένου να στηριχθεί και η επαγγελματική του κινητικότητα, η συμπερίληψη των γυναικών στην εργασιακή αγορά, αλλά και ευρύτερα η κοινωνική του ένταξη, ιδίω των μεταναστριών Νομίζω ένα από τα βασικά μηνύματα τη έκθεση αυτή είναι ότι στηρίζει τους στόχου τη Ευρώπη 2020 για την εκπαίδευση και την παιδεία, ιδίω τον πρωταρχικό στόχο ώστε να καταπολεμηθεί η εγκατάλειψη του σχολείου, τη πρώιμη εγκατάλειψη του σχολείου. Ο συνάδελφο αναφέρθηκε σε συγκεκριμένε συστάσει που προέκυψαν από το Ευρωπαϊκό ε, Εξάμεινο. Όλα αυτά τα μηνύματα του σχεδίου έκθεση απηχούν τι προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ρόλο τη εκπαίδευση και της κατάρτισης, όπως ε, αναφέρονται και στην ανακοίνωση που εγκρίθηκε τον ε, Νοέμβριο του 2012, πρόσφατα δηλαδή, ώστε να στηρίξουμε την εκπαίδευση και την βελτίωση των δεξιοτήτων για καλύτερα οικονομικά και κοινωνικά αποτελέσματα. Οι προτεραιότητε αυτέ την ε, περασμένη Παρασκευή εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Υπουργών Παιδείας και Εκπαίδευσης στα συμπεράσματά τους οι προτεραιότητε αυτές λοιπόν στον επανασχεδιασμό τη εκπαιδευτική μα πολιτική είναι απαραίτητε προκειμένου να βελτιωθεί το εκπαιδευτικό σύστημα και να καλύπτονται οι ανάγκες της εργασιακή αγοράς να ε, βρίσκονται οι απαραίτητε ικανότητε και δεξιότητε εκεί που αναζητούνται να αντλήσουμε τα απαραίτητα ωφέλη από την διαβίου μάθηση και με τη στήριξη των κατάλληλων φορέων. Θα πρέπει να υπάρξει αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και να στηριχθεί το σχετικό σύστημα αυτό, είτε πρόκειται για επίσημα είτε για άτιμα συστήματα. Επίση, η βελτίωση των βασικών δεξιοτήτων για νεαρού ανθρώπου και ενηλίκου, χωρί επαγγελματικέ δεξιότητε, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών. Πρόσβαση σε υψηλή ποιότητας φροντίδα για τα παιδιά. Οι γλωσσικές δεξιότητες προκειμένου να υπάρχει καλύτερη ένταξη στην κοινωνία γενικότητα και συγκεκριμένα στην ε, αγορά εργασίας. Η ανακοίνωση Thinking Education, δηλαδή η νέα αντίληψη για την εκπαίδευση, νομίζω σωστά συμπεριλαμβάνουν όλε αυτέ τι διαστάσει, ακόμα και τι τεχνολογικέ και επικοινωνιακέ δυνατότητε, στηρίζοντα την μάθηση, άτυπη και επίσημη αλλά και τη δυνατότητα να υπερβεί κάποιος, ε, κανείς τους φραγμούς που ακόμη συναντούν οι γυναίκες στην κινητικότητά τους. Τέλος, ήθελα να καλωσορίσω την έκκληση της έκθεσης να στηριχθεί το πρόγραμμα Εράσμους και να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να θυμίσω ότι το μελλοντικό Εράσμους for All ε, το πρόγραμμα αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συμπεριλαμβάνει μεγαλύτερη έμφαση στην κινητικότητα και τους πόρους για την ε, μαθησιακή κινητικότητα, όχι μόνο στην ανώτερη εκπαίδευση, αλλά στην ε, διαβίωση, κατάρτιση και μάθηση, με ανάλογα προγράμματα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο και πάλι στην κυρία Ραντσούλη για να κλείσουμε τη συζήτηση αλλά αν μπορέσετε να είστε σύντομοι στι ε, τελικέ σα παρατηρήσει, διότι θα πρέπει να προχωρήσουμε έτσι, να το ξανασυζητήσουμε το θέμα όταν φτάσουμε στι συμβαστικέ τοπολογίε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι συντομότατη, διότι δεν έχω σημαντικότατε παρατηρήσει. Απλώ θα πρέπει να απαντήσω, διότι κάποιοι συνάδελφοι στάθηκαν σε κάποιε επικρίσει και ήθελα να δώσω κάποια απάντηση. Στη συνάδελφο Τζούμπερ να πω δεν, ότι δεν πιστεύω ο υποχρεωτικό χαρακτήρα του να γίνουν με στατιστικά στοιχεία διαφανή τα μισθολόγια ανδρών και γυναικών ε, δεν είναι το κατάλληλο μέσο για να φτάσουμε στην μισθολογική ισότητα. Αντιθέτως, ε, με τη δουλειά μας στην καθημερινότητα θα πρέπει να υπάρξει ριζική αλλαγή στην οτροπία και την επαγγελματική κουλτούρα και ίσως έτσι να πετύχουμε ε, να πετύχουμε την τόσο την επιζητούμενη, την ποθητή αυτή επαγγελματική ισότητα. Στη συνάδελφο Κλειβέτη τώρα. Να πω κάτι για τις ιατρικές ε, υπευθύνου. Τις γυναίκες και την ε, θεμητή της ανησυχία ότι μπορεί να δημιουργείται έτσι έλλειμμα απαραίτητων εργαζομένων στη χώρα προέλευσης. Να θυμίσω ότι αναφερόμαστε στην έκθεση για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων. Από τη χώρα τη συναδέλφου μου, τη Ρουμανία, υπήρχε έντονη ε, κίνηση από τον παριατρικό κλάδο με πάρα πολλέ νοσοκόμε. Οπότε εδώ φαίνεται, αν ανησυχούμε ή όχι για τους ασθενείς, να αναγνωριστούν τα επαγγελματικά τους προσόντα για να μπορέσουν οι γυναίκες αυτές να αναζητήσουν δουλειά αλλού. Εάν ισχύει αυτό λοιπόν για τις νοσοκόμεους, ισχύει και για τις ε, γιατρούς. Εάν μια γυναίκα, γιατρός, αφού σπουδάσει, αναγκάζεται να φύγει σε άλλη χώρα, προφανώς το κάνει γιατί δεν έχει δουλειά στη χώρα της. Τώρα, το να προλάβουμε τέτοιε καταστάσεις είναι διακριτική μεταχείριση για αυτό το είδος του επαγγελματικού κλάδους. Τώρα, όπω σωστά αναφέρατε στην τροπολογία τη συναδελφού, βεβαίω πρέπει να βρεθούν λύσει αντιστάθμιση. Αντιστάθμιση για αυτό το πλήγμα που μπορεί να επιφερθεί. Αυτό ε, θα μπορούσαμε να το επεξεργαστούμε, σκεπτόμενοι την ε, κατάρτιση, την προώθηση επιπλέον προσωπικού, πρόσθετου προσωπικού. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για αυτά τα σχόλια. Σε 15 δευτερόλεπτα θα ξεκινήσουμε τη ψηφοφορία. Πρέπει και εγώ να δω τον κατάλογο ψηφοφοριών. Σε 15 δευτερόλεπτα ξεκινάμε. Okay, uh, Καλώς ξεκινούμε την ψηφοφορία. Σημείο 13. Ενσωμάτωση εφαρμογή οδηγίας του, του Συμβουλίου. Κυρία Γκουρμάη, θέλετε το λόγο. Παρακαλώ καθίστε όλοι και όλες και μην ε, φωνασκείτε. Η κυρία Γκουρμάη. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητές συνάδελφοι, Θέλω να σας υπενθυμίσω πόσο σημαντική είναι αυτή η οδηγία, η πρώτη ευρωπαϊκή οδηγία που ασχολείται με τις διακρίσεις ε, βάση φύλου εκτός αγοράς εργασίας. Είναι ζωτική σημασία η ενσωμάτωσή της στις εθνικές νομοθεσίες και η απαρέγκλητη τήρησή της, ειδικότερα σήμερα που ε, χρησιμοποιείται η κρίση ως πρόσχημα για να καθυστερείται ή να ακυρώνεται η χρηματοδότηση ε, για την ενίσχυση της ισότητας των φύλων. Έχουμε τις διατάξεις ε, που είναι αρκετά ασαφείς για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Είναι δυσνόητες αυτές οι διατάξεις για τους Ευρωπαίους πολίτες. Γι' αυτό καλό για περισσότερη διαφάνεια στην έκθεσή μου ως προς τις ασφαλιστικές εταιρείες, ούτως ώστε να μην υπάρχουν διακρίσεις στην ασφάλιση. Θα πρέπει η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη όλα αυτά να τα πάρουν πολύ στα σοβαρά και ελπίζω να, είμαι, να μπορέσω να στηριχθώ στη στήριξή σας και στην υπερψήφιση ε, της έκθεσης αυτής. Ε, βεβαίως, αν υπάρξουν προφορικές τροπολογίες, τι βλέπουμε, ο πρόεδρος θα ε, οργανώσει πολύ σωστά τη συζήτηση. Τροπολογία 8. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 9. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 11 υπέρ. 10 με συγχωρείτε υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε, να επαληθεύσουμε ηλεκτρονικώς. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Α, ε, ξεκινάει η ψηφοφορία για τροπολογία υπαριθμών 11. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Επομένως η 12 καταπίπτει. Πάμε στη 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Και εδώ να επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Ξεκινάει η ψηφοφορία για την 13. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές, να νομίζω ότι εγκρίνεται. Θέλετε να επαληθεύσουμε ηλεκτρονικός καλώς. Ξεκινάει η ψηφοφορία για τη 15. Τροπολογία 15. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία. Επομένως, 16, 17 και προφορική τροπολογία και οι τρεις καταπίπτουν. Πάμε στη συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 2. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Θέλετε να υπαρθέψουμε ηλεκτρονικώς. Ξεκινάει η ψηφοφορία για τη συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 3. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές ήταν πολύ ασαφές. Θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικώς. Τροπολογία 20 ξεκινάει η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Όχι, ήταν πολύ σαφές. Εγκρίνεται κατά κράτος θα έλεγα. 23 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά Αποχές. Απορρίπτεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 29 υπέρ. Θέλετε την 28 να την επαληθεύσουμε για της ηλεκτρονικής οδού. Ξεκινάει η ψηφοφορία για την 28. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 30. Υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ναι. Επαληθεύουμε την ε, τροπολογία 1, ξεκινάει η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σύνολο της νομοδότησης. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. εγκρίνεται. Σας ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. We done. go to the next... Τώρα προχωράμε στο επόμενο σημείο. Ατζέντα για παρκής, ασφαλής και βιώσιμες συντάξεις. Θα ήθελα η εισηγήτρια να λάβει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο λόγια για να ευχαριστήσω όλες τις συναδέλφους για τις συνεισφορές του την έκθεση αυτή. Λάβαμε 75 τροπολογίες, πολλές, ε, πραγματικά πολύ κοντινές τις ιδέες που περασπιστήκαμε στι εκθέσει αυτές, κάποιες καινούργιε. Σε κάθε περίπτωση προσπαθήσαμε να στηρίξουμε τις δύο βασικές προτεραιότητε του όλου αυτού εγχειρήματο. Πρώτον, την εξάλληψη όλων των μορφών ανισότητα ανδρών και γυναικών σε θέματα συνταξιοδότησης και σύνταξή, και έπειτα να εγγυηθούμε την ε, ε, βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων αυτό δείχνει ότι πολλές τροπολογίες που προέβλεπαν στη, προγράμματα στήριξης για μειονεκτούντες, ιδίως για άντρες και γυναίκες που πρέπει να ασχοληθούν με τα παιδιά τους ή άλλα μέλη της οικογένειας, αυτά θα πρέπει να υπολογιστούν με βάση τις κανονικές συντάξει και τα σχετικά δικαιώματα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία με την τροπολογία 24. Υπέρ, κατά, αποχέ, απορρίπτεται. 25. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 27. Υπέρ, κατά, αποχέ. εγκρίνεται. 26. Υπέρ,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 Είναι τη φορά, εγκρίνεται, αλλά ήταν ε, δύσκολο το αποτέλεσμα γιατί πολύ σηκώσατε τα χέρια σας. Θα κοιτάζω προσεκτικότερα. Περνάμε στην τροπολογία υπεριθμών 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 34, 35. 35 υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. Να κάνουμε έλεγχο για την 35. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Ας κάνουμε έλεγχο για την 39. Άρχεται η ψηφοφορία. 39. 39. Πέρας. Εγκρίνεται. 40 κατά τμήματα ψηφοφορίες. Ξεχωριστή μάλλον. Ναι, κατά τμήματα ψηφοφορίες. Πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Υπέρ 44 υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω ότι απορρίφθηκε. 46 υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος. Ε, ελέγχουμε την 46. 46, κάνουμε έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία. να ψηφίζει ο καθένας τον εαυτό του, κύριε Ταραμπέλα. Πέρας, απορρίπτεται. Τροπολογία 45. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 47. 47 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 49 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 53 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 50 παρομοιότυπη από την 51 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 52 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 60 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίφθηκε. 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 64 υπέρ κατά αποχές Νομίζω θα μπορούσαμε να ελέγξουμε για την 64. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται, τώρα η ψηφοφορία. Πέρας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 αποχές εγκρίνεται. 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πρώτη τροπολογία υπέρ κατά αποχές νομίζω να ελέγξουμε για την πρώτη τροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία υπαριθμών 1.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 Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στην εισηγητρία. Προχωράμε τώρα στο επόμενο σημείο, την κατάσταση των γυναικών στη Βόρεια Αφρική. Θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω θερμά τους και τις συναδέλφους σκιώδης εισηγητές και εισηγήτρες και τον Πρόεδρο για την δουλειά σας με τις τροπολογίες, όλους τους συναδέλφους που πρότειναν κέρυες τροπολογίες στην εκθεσή μου. Νομίζω ότι εδώ και ελπίζω να υπάρξει ευρεία υπερψήφιση, έκανα ό,τι μπορούσα ώστε να υπάρξει η σωστή συμφελίωση όλων των τροπολογιών, όλων των πολιτικών προελεύσεων. Ήταν σημαντικό να στείλουμε ένα χειρό μήνυμα προς τις γυναίκες αυτών των τεσσάρων χωρών της Βορειοαφρικής, οι οποίες ε, ζουν στην ε, κατάσταση αυτή των ευαίσθητων ε, διαδικασιών με πολλές ε, δυσκολίες και ε, αναταράξεις στην ανθρωπή των χωρών τους. Ένα μήνυμα και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση όμως αυτόν και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι θα πρέπει οι γυναίκες αυτές να ληφθούν υπόψη στη νέα εταιρική σχέση την Ευρωπαϊκή με τη Μεσόγειο στα προγράμματα που έχουμε καταρτήσει μέσω της εταιρική αυτής σχέσης. Πιο συγκεκριμένα, νομίζω ρόλος της έκθεσης αυτής είναι να τονίσει την πρωταγωνιστική δράση των γυναικών σε χώρες αυτές, όπως η Λιβύη. Με την Αραβική Άνοιξη φάνηκε και η διάσταση αυτή. Θα πρέπει αυτό να αναγνωριστεί λοιπόν στα, στην φάση της συνταγματικής διαδικασίας της πολιτικής αυτής ε, αναμόρφωσης και να προστατευτούν τα δικαιώματα των γυναικών αυτών, της εκπαίδευσή τους, της ε, επαγγελματικής τους ανέλυξης και της συμμετοχής τους στη λήψη πολιτικών αποφάσεων. Αισθάνομαι ότι εμείς εκπροσωπούμε σήμερα τόσες γυναίκες που ήδη έχουμε ακούσει και στο Ευρωκοινοβούλιο και επισκεπτόμενες αυτές τις τέρες, τέσσερις χώρες τους προηγούμενους μήνες γυναίκες που μας ζήτησαν να μιλήσουμε εκ μέρους τους, να δανείσουν, ζήτησαν να, μας, ε, να τους δανείσουμε τη φωνή μας, όχι να μιλήσουμε εκ μέρους τους, ε, να τις υποκαταστήσουμε μάλλον, αλλά να μιλήσουμε για το ρόλο τους στην δημοκρατική αυτή διαδικασία, τη γέννηση της δημοκρατίας και τη συμβολή τους, την πολιτική τους συμβολή. Είναι σημαντικό αυτό λοιπόν και Σημαντικό είναι και η Ευρωμεσογειακή Συνέλευση κάθε χρόνο μία συνεδρία, μία σύνοδο να την αφιερώνει στην κατάσταση των γυναικών και να τους δίνει ακριβώς το, ρόλο, το λόγο, να τους δίνει την ευκαιρία να εκφράσουν τη φωνή τους. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Θα αρχίσουμε τώρα την ψηφοφορία. Αρχίζουμε με την συμβιβαστική απολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 51 τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 52. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άρα λοιπόν, η άλλη Τροπολογία 50. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 53. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 57. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεν ψηφίζουμε για τροπολογία 56. Πάμε στην 58. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν κρίνεται. Βλέπω ότι Κάποιοι είστε μπερδεμένοι, είναι όλα σαφή. Βρίσκομαι εδώ για να σας καθοδηγήσω. Αν κάτι δεν καταλαβαίνετε, σηκώστε το χέρι, πείτε πρόεδρε κάνεις λάθος. ωραία, είμαστε εντάξει. Τώρα, τροπολογία 59, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 60, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Συμβασμός 2, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 68 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ηλεκτρονικά για την 68 άρχεται η ψηφοφορία. 68. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 78. Υπέρ. Υπέρ, κατά, αποχές. Θα το κοιτάξουμε ηλεκτρονικά. Την 78. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 78. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 79. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 6. Υπέρ. Κατά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 Άρα λοιπόν τώρα ψηφίζουμε για την συμβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άρα καταπίπτουν τώρα πολλές τροπολογίες και προχωρούμε στην 93. Όχι, 96, διότι 93 εγκρίθηκε. Ψηφίζουμε για την 96 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 103. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 110. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 111. Υπέρ, κατά, αποχές θα το κοιτάξουμε ηλεκτρονικά. Για την 111 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τώρα, συνολική τροπολογία της κυρίας Κράτσα, ε, προφορική τροπολογία, υπάρχουν αντιρρήσεις. Να ψηφίσουμε λοιπόν τροπολογία 112 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 113 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 114 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 115 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 116 υπέρ, κατά, αποχές, θα το κοιτάξουμε ηλεκτρονικά. 116. Άρχεται η ψηφοφορία για την 116. Πέρας. Εγκρίνεται. 117. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άρα οι άλλες τρεις καταπίπτουν. 119. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 120 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 121 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 122 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 123 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 124 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 125 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 126 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άρα 130 καταπίπτει. 127 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 128 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άρα οι επόμενε 7 καταπίπτουν. Συμβιβαστική 10 υπέρ. Κατά. απόχέ, εγκρίνεται. 136 υπέρ. Κατά. απόχέ, εγκρίνεται. 137 υπέρ. Κατά. απόχέ, εγκρίνεται. 2 ΔΕΒΕ 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 138 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 139 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 140 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 141 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρα 54 καταπίπτει. 142 τώρα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 146 τώρα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 147 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 148 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 150 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεβε 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεβε 6 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ο λόγος που είμαι τόσο γρήγορος είναι ότι επειδή βλέπω ότι όλοι σηκώνετε τα χέρια σας στην αρχή. Οπότε προχωράω λοιπόν. Προφορική τροπολογία 151. Υπάρχουν αντιρρήσεις για την προφορική τροπολογία. Ψηφίζουμε λοιπόν 151 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 152 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 153 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 154 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 155 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Κοιτάζουμε ηλεκτρονικά την 155. Άρχεται η ψηφοφορία για την 155. Πέρας. Απορρίπτεται. 156, προφορική τροπολογία. Υπάρχουν αντιρρήσεις για την προφορική. Όχι, άρα λοιπόν ψηφίζουμε για την 156. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 157. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 157. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 157. Πέρας. Απορρίπτεται. 158 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύε 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 159 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 160 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 161 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 162 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 163 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 164 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 165 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 166 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 167 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 168 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 169 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 170 προφορική τροπολογία. Συμφωνείτε όλοι. Ψηφίζουμε λοιπόν για την 170. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 171. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τέσσερα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μπορούμε να... Όχι, δεν μπορούμε, ναι, πρόεδρος, να τις ψηφίσουμε συνολικά. Συγγνώμη. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικά για την 7 άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 7. Πέρας. Εγκρίνεται.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 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να κοιτάξουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 16. Άρχεται η ψηφοφορία. 16. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές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 30 υπέρ κατά αποχές θα το κοιτάξουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 30. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται με μία ψήφο διαφορά. 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 29. Υπέρ. Κατά αποχές, κοιτάζουμε ηλεκτρονικά την 29. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 28 και 31 είναι ίδιες υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Τροπολογία 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται νομίζω. Θα κοιτάξουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 32. Άρχεται η ψηφοφορία για την 32. Πέρας. Απορρίπτεται. Με μία μόνο ψήφο. 33 υπέρ, κατά. Ξανά από την αρχή. 33 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 35 τώρα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άρα 37 καταπίπτει. Προχωράμε λοιπόν στην 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Θα κοιτάξουμε ηλεκτρονικά 38. Άρχεται η ψηφορία για την 38. Πέρας. Εγκρίνεται. 39. Υπέρ. Κατά. Από την αρχή. Υπέρ. Κατά. Θα κοιτάξουμε ηλεκτρονικά γιατί είναι 39. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. Σαφέστατα. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συνολικά η έκθεση. Άρχεται η ψηφοφορία. Μας λείπει ένας πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια. We now go to the last... Πάμε στην τελευταία ψηφοφορία. Αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης στην ισότητα των φίλων και στα δικαιώματα της γυναίκας. Θέλει το λόγο η συγγετρία. Δύο λόγια, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω μόνο τους συναδέλφους, τους σκιώδης εισηγητές από όλες τις πολιτικές ομάδες, οι οποίοι συνέβαλαν τα μάλα στη δημιουργία συμβιβαστικών λύσεων στο βαθμό του δυνατού για την έκθεση αυτή. Τους ευχαριστώ όλους ειλικρινά. Πρόκειται για συλλογική δουλειά οφείλω να σας πω ότι με χαρά θα επανεξετάσουμε το θέμα αυτό για την, ε, στις 7 Μαρτίου. Και εκεί θα έχουμε και πολύ ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις για αυτά τα τόσο καθοριστικά προβλήματα. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ καθίστε. Γιατί θα ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 7. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16. Ψηφοφορία κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται, νομίζω. Επαληθεύουμε ε, δια της ηλεκτρονικής οδού το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας υπαριθμών 16 μάλλον. Άρχεται η ψηφοφορία. Κάποιος λείπει. Απορρίπτεται. 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεν μπορούμε να τα ψηφίσουμε όλα μαζί. Χίδιν. Ίσως αργότερα, αλλά όχι τώρα. Όχι εδώ. 62. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 64 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Απασχόληση 1 πρώτο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 65. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται της Επιτροπής Απασχόλησης το 8 υπέρ. Πρώτο τμήμα. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 8, υπέρ. Οκτώ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην εννέα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 73 ψηφοφορία κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται. 74 ε, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ εγκρίνεται. 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Όχι. Ελέγχουμε ηλεκτρονικός. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Τροπολογία 83. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 9 της Επιτροπής Απασχόλησης. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 85 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 86 της Επιτροπής Απασχόλησης και 10. Ίδιες είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 87 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 90 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 88 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 89 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε δια της ηλεκτρονικής οδού την 89 ξεκινάει ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται με διαφορά μίας ψήφου. Τροπολογία 91 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 92 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 93 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 94 υπέρ αποχές, λέει ο πρόεδρος, κατά αποχές εγκρίνεται. 95 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 96 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 97 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 98 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 99 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 31 της Επιτροπής Απασχόλησης. Ένα τμήμα μόνο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συγγνώμη. Δεν έπρεπε να ψηφίσουμε την 31 της Επιτροπής Απασχόλησης γιατί έχει ήδη καταπέσει. Πάμε στην τροπολογία 100 και την 21 της Επιτροπής Απασχόλησης. Είναι ίδιες. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. να ελέγξουμε για της ηλεκτρονικής οδού την 104. Άμα το ζητάει κάποιος, πάντοτε εγώ το εκχωρώ. Ε, το κάνω. Λοιπόν, ξεκινάει η ψηφοφορία ηλεκτρονική για την 104. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 107. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 108 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ήταν πολύ ασαφές. Ποιος είναι υπέρ της 108. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Την 34 την ψηφίσαμε της Επιτροπής Απασχόλησης 109. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 της Επιτροπής Απασχόλησης. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφοφορία κατά τμήματα για την 113. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά, αποχές, νομίζω ότι απορρίπτεται. Το ελέγχουμε, το επαληθεύουμε. 113. Κάποιος το ζήτησε, όχι, τότε απορρίπτεται. Συμβαστική υπαριθμό 15. Αν δεν θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση να μην λέτε τίποτα. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 32 της Επιτροπής Απασχόλησης. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 16 συμβιβαστική υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 120 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 4 της Επιτροπής Απασχόλησης. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 122 τροπολογία. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 123 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 124 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 128 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 129 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 130 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 131 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 132 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 133 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 135 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 134 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 137 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 138 και 139 είναι ίδιες, ταυτόσιμες ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 140 υπέρ. Κατά άποχες εγκρίνεται. 33 της Επιτροπής Απασχόλησης. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 141 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 142 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 19 συμβιβαστική υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Πάμε λοιπόν στην 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μαζί, από 145 μέχρι 149, δεν θέλετε. Εντάξει, ξεχωριστά. Την 145, ποιος είναι υπέρ. Κατά να την επαληθεύσουμε. Την ψηφοφορία για την 145. Ξεκινάει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Ούτε τώρα τις υπόλοιπες τρεις μαζί. Εντάξει, τη 13 τότε. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Την 16 πάλι της Επιτροπής Απασχόλησης. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 146 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 148 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 149 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 155 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 21 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 152. Ψηφοφορία κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα της 152. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 156. Ποιος είναι υπέρ. Μαζί την 156 με... Δεν θέλετε. Εντάξει, δεν θέλετε. Στην 156 λοιπόν πάμε. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ξανά υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 157 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 158 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 160 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 22 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 163 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 164 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 165 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 168 υπέρ κατά αποχές Συγγνώμη, είναι προφορική τροπολογία. Υπάρχουν αντιρρήσει στην προφορική τροπολογία. Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν την 168. Υπέρ. Κατά άποχες εγκρίνεται. Τρία. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 29. Υπέρ. Κατά πρέπει να την ελέγξουμε την 29. Εξεκινάει ε, η ηλεκτρονική ψηφοφορία για επαλήθευση. Πέρας. Δεν είδα καθόλου χέρια να σηκώνονται, γι' αυτό το ζήτησα. Θα πρέπει να βρούμε και διαφορετικές λύσεις. Δεν βλέπω τόσο συντονιστές. Μπορώ να προσπαθώ να βλέπω γύρω-γύρω. 174 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 24 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 170 υπέρ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 171 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 172 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 176 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 177 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται.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 αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές θα πρέπει να ψηφίσουμε για τη 10 Πέρας. Εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμμεμπαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 23 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά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 47-48 πανομοιότυπες υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 49 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 50 υπέρ, κατά, εγκρίνεται νομίζω, 50, άρχεται η ψηφοφορία για την 50, πέρας και εγκρίνεται. 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Όχι, όχι, δεν γίνεται. 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, εγκρίνεται 55, 56 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τέλος, ηλεκτρονική τελική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία, ευθύς αμέσως, πέρας, εγκρίνεται με σαφή διαφορά. Σας ευχαριστούμε, συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Τελικό σημείο, σημείο 17, συνεδρίαση, επόμενη συνεδρίαση, 20 Μαρτίου 2013, από τις 9 έως τις 6.30. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας.